Περνάμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξη, που είναι δηλώσει του Συμβουλίου και τη Επιτροπή για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 20 και 21 Μαρτίου 2014. Και θα δώσω το λόγο στον κύριο Κούρκουλε, μέρο του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, ε, το Ενό Συνέδριο παραδοσιακά αφιερώνεται ε, στην οικονομική πολιτική. Αλλά ε, πριν εξετάσουμε την οικονομική ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου τη επόμενη εβδομάδα, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τα υπόλοιπα σημεία στην ημερήσια διάταξη. Τα διεθνή γεγονότα, άλλη μια φορά, επευλήθησαν στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η κατάσταση στην Ουκρανία είναι το πρώτο μέλημά μας και ήταν βεβαίως και ο λόγος για την, συνάντηση, την έκτακτη συνάντηση αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της προηγούμενης εβδομάδας. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα για το θέμα αυτό, εφόσον αποτελεί θέμα της ε, συζήτησης που θα ακολουθήσει. Απλώς ε, θα πω ότι είναι πολύ πιθανόν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας να επανέλθει στο θέμα αυτό. Επίσης για τις εξωτερικές σχέσεις, ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου θα συζητήσει και τη διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής, όπου θα συγκεντρωθούν, όπως γνωρίζετε, περίπου 100 επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων στις Βρυξέλλες στις 2 και 3 Απριλίου. Ε, Όπω είπα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου παραδοσιακά εστιάζεται στην οικονομική και κοινωνική πολιτική. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποφάσισε να διαρθρώσει την συζήτηση γύρω από τρία βασικά ζητήματα τη στρατηγική μα για την ανάπτυξη την ε, ε, απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα. Το πρώτον θα είναι το ευρωπαϊκό εξάμεινο, δεύτερον η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και τρίτον το κλίμα και η ενέργεια. Αυτά είναι τα τρία βασικά θέματα. Και δεν είναι τυχαία η σειρά των θεμάτων, να αλληλοσυνδέονται αυτά τα θέματα. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αποτελεί το εργαλείο για την παρακολούθηση τη υλοποίηση τη στρατηγική για την Ευρώπη 2020, ενώ η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, το κλίμα και η ενέργεια είναι δύο από, τα, από τι συνιστώσει. Δεν μπορεί να υπάρξει βιομηχανική ανταγωνιστικότητα χωρί συνεκτική πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια και αντιστρόφω. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ολοκληρώσει την πρώτη φάση Ήδη το Δεκέμβριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε στοιχεία καθοδήγησης για τις προτεραιότητες πολιτικής για τα επόμενα χρόνια και αυτό δείχνει και τη σημασία που έχει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Την επόμενη εβδομάδα θα εξετάσουμε ε, την υλοποίηση των συστάσεων ειδικά για κάθε χώρα για το 2013 και θα δώσει καθοδήγηση για την περαιτέρω εργασία για, για τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλησης και τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης όσον αφορά την οικονομική και κοινωνική διάσταση. Εποφελούμε τις ευκαιρίες σήμερα για να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το σημαντικό έργο που έχει αναλάβει για, διάφορα, για διάφορες πτυχές του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πλησιάζουμε το τέλος ενός οικονομικού κύκλου. Οι συνέπειες της κρίσης είναι ακόμη αισθητέ. Η ανάπτυξη ε, δεν είναι ομοιογενής και είναι και εύθραυστη. Όμως μάλλον έχουμε αφήσει πίσω μας τα χειρότερα. Και αυτό είναι ένας λόγος ε, που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξετάσει την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής του 2020. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, θα φροντίσει να γίνει μια αναθεώρηση της στρατηγικής ε, εγκαίρως ε, πριν από το Ερεινό Συμβούλιο Κορυφής. Η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή ανταγωνιστική βάση. Η βελτίωση τη ανταγωνιστικότητά μα είναι θεμελιώδου χαρακτήρα. Είναι βασικό συστατικό για να διασφαλίσουμε μια ε, βιώσιμη ανάκαμψη των οικονομιών μα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει πώ μπορούμε να επιτύχουμε ε, ισχυρή βιομηχανική βάση στην Ευρώπη. Θα εξετάσει το πώ μπορούμε να ενισχύσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο και την εσωτερική αγορά και όχι μόνο αυτό. Οι ηγέτες της Ευρώπης ε, θα προσπαθήσουν να υποστηρίξουν ε, την ε, ανταγωνιστικότητα ως τμήμα όλων των πολιτικών και να γίνεται μια συστηματική εξέταση όλων των πολιτικών ως προς την ανταγωνιστικότητα για να είναι σίγουρο ότι θα υλοποιηθούν αυτά τα στοιχεία που θα συζητηθούν. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα, θα φροντίσει να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη έχει πρόσβαση σε υψηλή κατάρτισης προσωπικό. Χρειαζόμαστε εξέταση των ε, ελλημάτων που υπάρχει σε τομεί όπω η μηχανική, τα μαθηματικά, για να καλυφθούν αυτές οι ελλείψεις. Επίσης θα κατευθυνθούμε προς τομείς υψηλής ανάπτυξης θα ε, εξετάσουμε ε, επίσης την προτεραιότητα στην ε, καινοτομία. Η ανταγωνιστικότητα είναι ζωτική σημασία και όταν εξετάζουμε τη βιομηχανία μας από την οπτική γωνία των διεθνών αγορών. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ένταξη των ευρωπαϊκών εταιριών σε αλυσίδες παγκόσμιας αξίας και να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας μέσω μιας φιλόδοξης ημερήσης διάταξης για το εμπόριο και την ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει μια πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα που θα είναι συνεκτική. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα κάνει λοιπόν μια πρώτη συζήτηση για ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα στην περίοδο από το 2020 έως το 2030. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται ότι θα ζητήσει μια συμφωνία αρκετά σύντομα ώστε να ληφθεί υπόψη το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε στη Βαρσοβία και τα διεθνή γεγονότα που θα ακολουθήσουν, η COP21 στο Παρίσι του χρόνου και μια φιλόδοξη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών μέχρι το 2030 είναι ένας τομέας ε, που θα πρέπει περαιτέρω να αναπτυχθεί στο ε, μέλλον. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, σημειώνει την πρόοδο που έγινε από την προηγούμενη συνάντησή του για την ενέργεια το Μάιο και η ολοκλήρωση της αγοράς μέχρι το 2014 και η ανάπτυξη αλληλοσυνδέσεων για να μην υπάρχει αποκλεισμός κάποιων κρατών μελών από τα ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου μέχρι το 2015 παραμένουν προτεραιότητα. Δεν χρειάζεται να τονίσω πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα και μάλιστα υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων στην Ουκρανία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εντοπίσει κάποιους τομείς όπου απαιτείται περαιτέρω εργασία για να καταλήξουμε σε αυτούς τους στόχους. Θα εξετάσει επίσης το πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα του υψηλού ενεργειακού κόστους. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, αναμένουμε ότι αυτό το, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα είναι ένα συμβούλιο που θα ασχοληθεί με τα οικονομικά θέματα ω συνήθω, αλλά πάντοτε προστίθενται και κάποια θέματα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξετάσει όλα αυτά τα θέματα παράλληλα με θέματα του πώ ε, ε, να επιτύχουμε ανάπτυξη απασχόληση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Όπως πολλές φορές έχουμε πει στη συζητήση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οικονομική και κοινωνική πολιτική αποτελεί ένα ισχυρό σημείο για την Ευρώπη. Μας δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη διεθνή σκηνή και μας δίνει τη δυνατότητα να παίξουμε ένα ηγετικό ρόλο παγκοσμίω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κούργουλα. Εκ μέρους της Επιτροπής ο Πρόεδρος Μπαρόζο έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, αγαπητά μέλη, είναι αυτονόητο ότι ε, τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα στην κρίση της Ουκρανίας. Είμαι σίγουρος ότι το Ευρωπαϊκό ε, Συμβούλιο θα ασχοληθεί επί μακρόν με αυτό το μεγάλο ζήτημα. Επειδή όμως θα το συζητήσουμε αργότερα το πρωί, θα επικεντρωθώ στα άλλα βασικά στοιχεία που θα απασχολήσουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα λάβει γνώση της προόδου που έχει επιτελεστεί σε σχέση με την αντιμετώπιση της οικονομικής ε, κρίσης και στα πλαίσια βεβαίως και της ε, αναδιάρθρωσης, των αναδιαρθρώσεων. Θα λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία για να ενισχύσουμε τις συγκεκριμένες μας δράσεις σε σχέση με το θέμα της ανεργίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίσης θα είναι το τελευταίο πριν από τις εκλογές και θα πρέπει να κρατήσει αυτή την όθηση ως προς το ευρωπαϊκό εξάμεινο και τα άλλα θέματα της ατζέντα. Εμείς έχουμε προβεί σε μία εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης και των μακροοικονομικών συνιστοσών. Μερικές εβδομάδες πριν στην Ολομέλεια είχαμε μία συζήτηση η οποία ε, οδήγησε σε ένα ψήφισμα για το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Υπήρξε μεγάλη σύγκληση ως προς τις προτεραιότητες όπως διαμορφώθηκαν. Όπως ξέρετε έχουμε αναθεωρήσει τις οικονομικές εκτιμήσεις. Θα έχουμε ε, μία, ένα δίκτυο ανάπτυξης 1,5% φέτος και 2% του χρόνου. Αυτό αποτελεί μία μικρή ε, πρόοδο. Η ανάπτυξη επανέρχεται στην Ευρώπη και αυτό αφορά και τα πιο ευάλωτα κράτη-μέλη. Η εγχώρια κατανάλωση θα επεκταθεί έτσι ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε στον εξωτερικό τομέα για την ανάκαμψή μας. Αυτό μας οδηγεί σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να επιτελεστούν για να επιτύχουμε την ανάπτυξη. Η ανταγωνιστικότητα είναι ένα μεγάλο θέμα σε πολλές ε, ε, χώρες, γι' αυτό η στρατηγική μας για το 2020 θα βελτιώσει τις προοπτικές ανάπτυξης για πολλές χώρες. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο για τους πολίτες, διότι η ανάπτυξη είναι πρόκριμα των θέσεων εργασίας, για την ε, αντιμετώπιση της ανεργίας. Κάτι το οποίο είναι μία από τις ε, ε, προτεραιότητές μας. Γι' αυτό θα θέλαμε να προωθήσουμε το Ταμείο για την Νεολαία και διοργανώνουμε μία διάσκεψη τον επόμενο μήνα στις Βρυξέλλες για να κρατήσουμε αυτή την ορμή, τη μεγάλη όθηση για την αντιμετώπιση της ανεργίας κυρίως των νέων. Η εμπιστοσύνη βασίζεται στην αξιοπιστία και η αξιοπιστία ε, βασίζεται στο να ανταποκριθούμε στις ε, υποχρεώσεις μας. Μετά από την απόφαση για την Τραπεζική Ένωση του 2012 θα πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις αγορές, κάτι το οποίο προωθούμε φέτος. Τώρα θα πρέπει να φτάσουμε και στο τελικό στοιχείο, δηλαδή στον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης προωθήσαμε την πρότασή μας στεναρά και το Συμβούλιο θα πρέπει να ανταποκριθεί έτσι ώστε να μας δώσει ορισμένα στοιχεία για να φτάσουμε σε διακυβερνητική συμφωνία. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Γι' αυτό η συνάντηση του Συμβουλίου σημαίνει ότι η διακυβερνητική θα πρέπει να έχει έναν ελάχιστο παρονομαστή Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια επιτάχυνση λειτουργίας των ε, ταμείων για να μπορέσουν να λειτουργήσουν από την πρώτη ημέρα και να υπάρχει αυτονομία ως προς το ευρωπαϊκό δίκαιο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, έτσι ώστε ο καθένας να ορίσει τα δικά του. Χτες στην ΕΚΟΦΗΝ δεν επιτελέστηκε πρόοδος σε σχέση με τον αντίστοιχο ρόλο του Συμβουλίου και της Επιτροπής και η Επιτροπή ασχολείται ως προς την συμμόρφωση του Συμβουλίου με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η Επιτροπή ε, συνεργάζεται μαζί σας για να φτάσουμε σε μία αίσια έκβαση κοντά στο αρχικό μας ε, πρόγραμμα. Ε, θεωρώντας ότι υπερέχει πάντα το κοινοτικό δίκαιο. Αγαπητά μέλη, θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα δεχτεί και την ανακοίνωση Επιτροπής για την βιομηχανική ανάκαμψη διότι πολύ είναι οι μοχλοί για να ε, ανακάμψει η βιομηχανία μας, αλλά βρίσκονται στο, σε εθνικό επίπεδο. Πολλές βιομηχανίες μας έχουν χάσει την ανταγωνιστικότητα και η έρευνα και η καινοτομία βρίσκονται αρκετά πίσω. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να ε, μπορέσουν να ανταποκριθούν οι ευρωπαϊκές ε, βιομηχανίες που έχουν μεγάλα προβλήματα προμήθειας ε, κεφαλαίων και εργατικού δυναμικού, εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Εμείς θα πρέπει να ορίσουμε κανόνες που να είναι φιλικοί προς το χρήστη, να έχουμε ευφυή δίκτυα και επενδύσεις για ε, τον ορίζοντα 2020. Επίσης θα πρέπει να ε, ορίσουμε μια ευφυή ε, βιομηχανία για τα επόμενα χρόνια χρηματοδότηση των ΜΜΕ, ε, βελτίωση των δεξιοτήτων, μείωση της γραφειοκρατίας και υποστήριξη της ε, διπλωματίας. Αυτό είναι το έργο μας, αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει επίσης να είναι αποφασιστικά, διότι πολλά ζητήματα θα πρέπει ε, να, μάλλον αφορούν τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να ανταποκριθούν τα κράτη-μέλη. Η αγορά εργασίας έτσι θα είναι αποτελεσματική και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Επίσης θα πρέπει να μειώσουμε το άχθος της ΜΜΕ και να ορίσουμε καλύτερο πλαίσιο επενδύσεων, διότι μόνο η τεχνολογική ανάπτυξη εγγυάται την ανταγωνιστικότητα τέλος θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα για να αρθούν τα προσκόμματα στην ολοκλήρωση της ενίας αγοράς που επιθυμούμε. Διότι αυτό είναι το πιο δύσκολο πρόβλημα, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την ψηφιακή αγορά και την ενέργεια. Θα πρέπει να φτάσουμε σε μια εσωτερική αγορά ενέργειας για να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας, όπως όρισε και το Συμβούλιο. Και αυτό βεβαίως θα συζητηθεί και ελπίζω να δοθεί ένα σαφές ε, μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το ίδιο ισχύει για την πολιτική μας ε, σε σχέση με τις αλλαγές του κλίματος μαζί με την ενέργεια. Αυτό θα συζητηθεί στο επόμενο ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μαζί με την Ουκρανία. Θα πρέπει να υπάρχει ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων για να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Η αύξηση της τιμής της ενέργειας είναι ανησυχητική για τις επιχειρήσεις. Επίσης, οι πράσινες τεχνολογίες είναι ζωτική σημασία για την εργασία και την ανάπτυξη, αν θέλουμε να υπάρχει ε, βιωσιμότητα. Επίσης, υπό το φως της κρίσης ε, της Ουκρανίας μην ξεχνάμε την εξάρτηση της Ευρώπης ε, από την ενέργεια. Μιλάμε για την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές. Ελπίζουμε αυτό το σχήμα να είναι εφικτό. Βρισκόμαστε σε καλό σημείο για να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων για τους κανόνες 2020 ε, και να κινηθούμε προς το 2030 το στρατηγικό πλαίσιο κλίματος και ενέργειας κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Ορίζει μείωση εκπομπών θερμοκηπίου της τάξης του μείω 40% μέχρι το 2030, συγκρίνοντας με το 1990. Επίσης, θεωρούμε ότι είναι εφικτό και αποδοτικό όπως δείχνει η έρευνά μας διότι το 40% είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για τους στόχους μας για το 2050. Επίσης θα πρέπει να ορίσουμε ένα στόχο για το 2030 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 27%. Θεωρούμε ότι οι ανανεώσιμες είναι ένα στοιχείο κλειδί γιατί ορίζουν και την ενεργειακή μας ασφάλεια θεωρούμε, δεν μπορούμε να ορίσουμε 28 διαφορετικούς ε, στόχους. Θα πρέπει να έχουμε μία άναντι προσέγγιση. Νομίζω ότι τα διδάγματα του παρελθόντος δείχνουν ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος και χρειαζόμαστε μία έναν ευφύ επιμερισμό εργασίας. Τα κράτη-μέλη θα ορίσουν τους στόχους ανανεώσιμων σε εθνικό επίπεδο και θα δεχτούμε και το ενεργειακό μείγμα που ορίζεται σε εθνικό επίπεδο. Όμως θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις ανανεώσιμες ε, θεωρώντας ότι παραμένουν μέσα στα πλαίσια της, ε, και των εθνικών επιδοτήσεων. Επίσης, θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσα ενός πλαίσιου ε, διακυβέρνησης. Θεωρούμε ότι η στρατηγική του 2020 δεν έχει δεσμευτικό στόχο. Εμείς θα, θα αναθεωρήσουμε το πλαίσιο μετά το 2014 πριν ορίσουμε τα επόμενα βήματα και θεωρούμε ήδη στη θητή αυτής της Επιτροπής να ορίσουμε το νέο πλαίσιο. Έχουμε ορίσει ένα πλαίσιο Τώρα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ανταποκριθούν καθώς και το Κοινοβούλιο. Το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας θα δώσει ένα σαφές μήνυμα σε σχέση με τη στρατηγική αυτή και θα ορίσουμε αυτή την μεγάλη όση που έχει αρχικά δοθεί. Αυτό είναι ύψης της σημασίας, διότι θέλουμε τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν σε αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο για μερικούς, αλλά θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να κρατήσουμε την ανταγωνιστικότητα σε πολύ υψηλό έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι να ανταποκριθούν. Δεν μπορούμε να κινηθούμε μόνοι μας. Πρέπει οι μείζονες οικονομίες να βρίσκονται στο πλευρό μας, καθώς και όλοι οι άλλοι εάν λάβουμε υπόψη τη διοργάνωση του Μπαν των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο φέτες. Δηλαδή το Σεπτέμβριο όταν μεταβούμε στη Νέα Υόρκη θα πρέπει να δείξουμε ότι η Ευρώπη ανταποκρίνεται στον ηγετικό της ρόλο. Δεν είναι ε, νωρίς, το 2030 είναι πολύ κοντά, δεν μπορούμε να κρατήσουμε στάση αναμονής. Θα πρέπει να δώσουμε στις επιχειρήσεις μας την ασφάλεια που επιθυμούν. Επίσης, θα πρέπει να ορίσουμε την ατζέντα μας σε διεθνές επίπεδο, αλλά ανταποκρινόμενοι στα ημέτερα. Πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά, διότι το απαιτούν οι περιστάσεις και θα πρέπει να δράσουμε από κοινού. Τα πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν ότι κάτι τέτοιο είναι ύψης της σημασίας τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κατέχουν ηγετικό ρόλο και εν ώψη των εκλογών και με βάση τις οικονομικές δυσχέρειες θα πρέπει να εργαστούμε στεναρά. Πολύ περισσότερο από το παρελθόν. Αυτό αναμένουν από μας οι πολίτες και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Μπαρόζο. Εκ μέρου ε, του ΕΛΚ ο κύριο Ντόλ. Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα τεταμένο διεθνέ πλαίσιο. Συρία, Αίγυπτο, Ουκρανία, Όλοι έχουμε στο μυαλό μας τις χώρες αυτές. Η σταθερότητα των γείτονων χωρών μας δείχνει πόσο εύθραυστο είναι το περιβάλλον μας και πόσο πρέπει να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να πάμε πιο μακριά και για να κρατήσουμε την ειρήνη. Στο συνέδριο του ΕΛΚΑ, ο Μπόνο, ο Ιρλαδός τραγουδιστής, μας έδωσε ένα μήνυμα γεμάτο κοινή λογική. Συμμερίζομαι τις διαπιστώσεις του. Μας είπε ότι η Ευρώπη είναι μια οικονομική οντότητα, υπάρχει, τώρα πρέπει να είναι παρούσα και να γίνει μια κοινωνική οντότητα. Ε, είναι αλήθεια. Η Ευρώπη πρέπει να είναι ενωμένη για να είναι δυνατή. Έτσι θα ακουστεί η φωνή μας ανά τον κόσμο. Οι αποφάσεις που θα λάβει το Ερνό Συμβούλιο όσον αφορά την ενέργεια, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα είναι ακριβώς αυτά που θα βοηθήσουν την Ευρώπη να, περάσει, να προχωρήσει και να φέρει σε πέρα στην αποστολή της. 28 χώρες δεν μπορεί να είναι όμοιροι προμηθευτών ενέργειας σε ασταθείς περιοχές του κόσμου που χρησιμοποιούν την ενέργεια ως οικονομικό όπλο. Δεν πρέπει να διατηρηθεί η εξάρτησή μας από εκεί. Οι πολίτες μας ανησυχούν. Οι πολίτες μας των ανατολικών χωρών, αναφέρομαι σε αυτές βέβαια, ανησυχούν πολύ. Υπάρχει ανεργία, υπάρχει πρόβλημα γενικά στην περιοχή τους. Αυτό είναι ένα θέμα που θα είναι κεντρικό στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Όλοι εδώ συμφωνούμε, αλλά χρειάζονται λύσεις για την απασχόληση που είναι όμως διαφορετικές μεταξύ μας. Χρησιμοποιούμε σλόγγαν, μιλάμε για λιτότητα και κάνουμε τον κόσμο να φοβάται. Ο Jean-Claude Juncker που είναι ο υποψήφιός μας για πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι οι άνεργοι στην Ευρώπη είναι το 21ο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 20 εκατομμύρια άνεργοι. Πρέπει λοιπόν να επικεντρώσουμε την, ε, τις προσπάθειές μας στην απασχόληση ακριβώς. Με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δώσαμε στην Ευρώπη ένα εργαλείο για να ενισχύσει την αξιοπιστία της. Αξιοπιστία απέναντι στους ε, επενδυτές πρώτα απ' όλα. Δεν είναι βέβαια αυτός σκοπός, αλλά πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει να υπάρχουν καλές επενδύσεις που θα στηρίξουν την ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό και οι στόχοι του ορίζοντα 2020 είναι πάρα πολύ σημαντικοί και θα βοηθήσουν τη βιομηχανική μας πολιτική. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία, χάρη στις μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις, αποτελούσε πάντα τη δύναμη της Ευρώπης. Η Ευρώπη έτσι εποφελήθηκε από την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Όμως επειδή δεν υπάρχει πραγματική φορολογική και κοινωνική εναρμόνιση, δυστυχώς φορκόπησαν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ανοίξτε τη εφημερίδα «Τα νέα της Αλσατίας» για παράδειγμα. Υπάρχουν δύο σελίδες που αναφέρονται σε πτωχεύσεις επιχειρήσεων. Μόνο εδώ στην Αλσατία, τη δικιά μου περιφέρεια. Είναι φοβερό. Μιλάμε για Απολύσει στις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά δεν μιλάμε για όλε αυτές τις εκατοντάδες επιχειρήσεις που εξαφανίζονται καθημερινά και αφήνουν βέβαια χιλιάδες άνεργους. Σήμερα έχουμε 20 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη που πρέπει να μπορούν να μιζάρουν στην ανταγωνιστικότητά τους, ένα ευνοϊκό περιβάλλον. Γιατί μόνο έτσι θα βοηθήσουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την απασχόληση αν η κάθε μικρομεσαία επιχείρηση προσλάμβανε έναν εργαζόμενο δεν θα υπήρχαν πια άνεργοι. Και θέλω τώρα να επανέλθω στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ορισμένοι πιστεύουν ότι χάνεται η κυριαρχία. Μα το αντίθετο συμβαίνει. Είναι κέρδος στην κυριαρχία. Γιατί με περισσότερη διαφάνεια, με επιμερισμένη εποπτεία, με συντονισμό ενισχύουμε την κυριαρχία, την ευρωπαϊκή κυριαρχία. Και το ευρωπαϊκό εξάμεινο ακριβώς είναι το οχυρό που θα μας βοηθήσει να αντισταθούμε στα επικίνδυνα συμβάντα που μπορεί να συμβαίνουν στον οικονομικό χώρο είναι κάτι πολύ βασικό για την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για την ειρήνη, για την ευημερία, για μια ενωμένη Ευρώπη, για μια Ευρώπη που προστατεύει. Ελπίζω 25 Μαΐου οι συμπολίτε μας να εκφραστούν και να πούνε ποια Ευρώπη θέλουν για αυτούς και για τα παιδιά τους. Για μένα η απάντηση είναι απλή. Χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη είναι η λύση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ντόλ. Ο συνάδελφος Βότσον έχει μια ερώτηση, αν συμφωνείτε να τη δεχτείτε. Κύριε Βότσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σίγουρα θα συμφωνήσετε κι εσείς. Πρέπει να συγχαρούμε τον κύριο Ντόλ που εξελέγει πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είπατε κι εσείς ότι το θέμα της Ουκρανίας δείχνει πόσο επικίνδυνο είναι να εξαρτώμεθα από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και για τη Γερμανία πολλά διακυδεύονται εδώ. Γιατί δεν στέλνετε στη Μόσχα λοιπόν την κυρία Μέρκελ για να συζητήσει μαζί τους για το θέμα της ενεργειακής πολιτικής και τις τιμέ και το αφήνετε στον Τζον Κέρι. Δεύτερον, αν επιταχύνουμε την αλλαγή από τα ορυκτά στην καθαρή ενέργεια, τότε κερδίζουμε και ανεξαρτησία από την Ρωσία, αλλά φέρουμε σε πέρα στις υποχρεώσεις μας σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές. Γιατί λοιπόν το ΕΛΚΑ εξακολουθεί να αντιτίθεται σε δεσμευτικούς στόχους όσον αφορά την πράσινη ενέργεια στην οποία αναφέρθηκε και μόλις πριν ο κύριος Μπαρόζο. Κύριε Ντόλ. Ναι, μα κύριε Βότσον. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για τα συγχαρητήρια. Ξέρετε, στην Αλσατία δεν λέμε ξύχανα συλληπιτήρια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ πολύ. Έπειτα. Γιατί να στείλω την κυρία Μέρκελ να μιλήσει με τους Ρώσους. Είμαι Ευρωπαίος. Η κυρία Μέρκελ καλά κάνει να έχει καλές σχέσεις με του Ρώσους, δεν έχω κανένα πρόβλημα, μπράβο της. Το ευρωπαϊκό εξάμεινο όμως, εδώ όλοι οι Ευρωπαίοι θα το διαπραγματευτούν και το θέμα της ενέργειας, γιατί μια χώρα, ακόμα και αν είναι η Γερμανία, δεν θα έχει το ίδιο βάρος που έχουμε όλοι μαζί για την ενεργειακή πολιτική. Αυτή είναι η πρώτη μου απάντηση. Έπειτα, αγαπητέ Βότσον, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι το ΕΛΚ είναι κατά του περιβάλλοντος. Όμως, μια στιγμή. Κι εγώ είμαι υπέρ του περιβάλλοντος, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε τις καλύτερες επιδόσεις. Είμαστε πολύ πιο μπροστά από τους υπόλοιπους. Και αν συνεχίσουμε, πρέπει να συνεχίσουμε. Αλλά αν οι άλλοι, η Κίνα και οι υπόλοιποι δεν μας ακολουθήσουν, τότε θα χάσουμε όλη μας την απασχόληση. Όλες οι θέσεις απασχόλησης θα χαθούν. Η Ευρώπη θα είναι η πιο καθαρή στον κόσμο, αλλά δεν θα έχει θέσεις απασχόλησης. Και το είδα και αυτό στη Γερμανία, στο Βερολίνο, που πήγα και μίλησα με τους επικεφαλείς μεγάλων επιχειρήσεων. Και υπάρχει ένας της Dissengruff, ο οποίος τι μου είπε, Εκτός μικροφώνου παρεμβάσεις. Εγώ θέλω να κρατήσουμε όλες τις θέσεις απασχόλησης που έχουμε. Να μην διακινδυνεύσουμε τις επιχειρήσεις μας εξαιτίας περιβαλλοντικών προβλημάτων. Είμαι κι εγώ ε, αγρότης και εγώ θέλω να προστατεύουμε το περιβάλλον, αλλά να το κάνουμε όλοι. Αν το κάνουμε όλοι, τότε θα το προστατεύσουμε καλύτερα. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Βόμποντα εκ μέρους ε, των ε, Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε περισσότερο ρεαλιστές. Ρεμπέκα, ησυχία παρακαλώ. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε περισσότερο ρεαλιστές. Οι πολίτες της Ευρώπης ε, συχνά νιώθουν απογοήτευση, μερικές φορές ε, και αηδία όταν σκέφτονται την, ε, την Ευρώπη. Ο Προεδρεύον του Συμβουλίου μίλησε για την καθοδήγηση που δίνει το Συμβούλιο. Μα πού είναι η καθοδήγηση του Συμβουλίου και πού μας οδηγεί. Δεν είναι καθόλου σαφές. Δεν είναι σαφές ούτε για τους πολίτες αλλά ούτε και για μας. Θα γίνει άλλο ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ως συνήθως, χωρίς καμιά αλλαγή και τα συμπεράσματα δεν θα έχουν τίποτα το καινούριο. Κάποιες, ε, κάποια συμπεράσματα χωρίς ε, ιδιαίτερο νόημα, κάποιες αόριστες ε, δεσμεύσεις αναζητώντας τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή υπάρχει ένα φιλελεύθερο νέφο που δεν αφήνει το Συμβούλιο να δει την πραγματικότητα. Παραδείγματο χάρη τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα που έχουμε στην Ευρώπη. Είμαστε μια από τι πιο πλούσιε υπείρου ή υπήρους, η πιο πλούσια ήπειρος, αλλά η κατανομή πλούτου και εισοδήματο γίνεται όλο και περισσότερο άνηση. Μιλήσατε για το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται. Γιατί φεύγουν τόσοι νέοι άνθρωποι από τη χώρα του, από την Ισπανία, από την Πορτογαλία, ακόμη και από τη Γαλλία. Υπάρχει κάποια έλλειψη ε, ισορροπίας μεταξύ των ε, προσόντων και ε, των θέσεων εργασίας και αυτό πρέπει να καλύψουμε. Αν κάνουμε μια σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν λέω ότι είναι όλα ρόδινα στις ΗΠΑ, αλλά είχαν ανάπτυξη 2,4% η ΕΠΑ, εμείς στην Ευρωζώνη 0,5%. Οι ΗΠΑ έχουν ανεργία 6,7%, η Ευρωζώνη σχεδόν διπλάσια ανεργία πληθωρισμός 1,7 στη ΣΥΠΑ, 0,8 στην, Ευρω... στην Ευρωζώνη. Ίσως ε, ο αποπληθωρισμός είναι το πρόβλημα και δεν κάνουμε τίποτα για να το αντιμετωπίσουμε. Τον Ιανουάριο ε, 11% το Ιανουάριο του 2012, το ίδιο το 2013. Πού είναι η πρόοδος στην οποία αναφέρεται και το ΑΕΠ πέρυσι παρουσίασε αύξηση 0,1%. Πού βρίσκεται η, ανάπτυξη. Μιλάμε για τους νέους που είναι καινοτόμοι, που είναι ερευνητές, που θέλουν να ξεκινήσουν με νέες εταιρείε. Τι κάνει όμως το Συμβούλιο για να μην έχουμε διαρροή εγκεφάλων. Το βλέπουμε στην Ευρώπη σήμερα, φεύγουν ε, οι νέοι, έχουμε διαρροή εγκεφάλων και δεν κάνουμε τίποτα για να κρατήσουμε τους νέους στην Ευρώπη, να τους δώσουμε μια δουλειά. Και η Επιτροπή και το Συμβούλιο αποτυγχάνουν παταγωδώς σε αυτό. Πρέπει να έχουμε ένα όραμα για το πώς θέλουμε να αναπτυχθεί η Ευρώπη, κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Φοροδιαφυγή. Στη Γερμανία και μόνο τώρα δικάζεται ένα συγκεκριμένο άτομο και αυτός ο ένας και μόνος άνθρωπος φαίνεται να δικάζεται για φοροδιαφυγή πάνω από 20 εκατομμύρια λόγω κερδοσκοπικών πράξεων στην Ελβετία. Μπορεί και 27 εκατομμύρια, εν πάση περιπτώσει πάνω από 20 σίγουρα. Ένας άνθρωπος μόνο που αυτή τη στιγμή δικάζεται. Τι κάνει το Συμβούλιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής δύο χώρε ακόμη αρνούνται να λάβουν μέτρα κατά της φοροδιαφυγής. Τι κάνετε γι' αυτό. Δεν υπάρχει λοιπόν θάρρος, δεν υπάρχει όραμα, δεν υπάρχει καθοδήγηση. Ότι είναι απογοητευμένοι οι πολίτε είναι αλήθεια και αυτός είναι ο λόγος που μπορεί να έχει και κάποια επιτυχία ο κύριο Φαράτζ. Όχι γιατί έχει απαντήσει, απαντήσει δεν έχει. Αλλά όταν αποτυγχάνει η πολιτική, οι λαϊκιστές, ακόμη και αν δεν έχουν απαντήσεις, μπορεί να, έχουν, να κερδίζουν ε, κάποιο πεδίο θυμάμαι τον Σάμιουλ Μπέκετ με αυτά που γίνεται τώρα στην Ευρώπη που έλεγε ας ξαναπροσπαθήσουμε, ας αποτύχουμε, αλλά ας αποτύχουμε καλύτερα. Δεν έχουμε χρόνο όμως για να αποτύχουμε καλύτερα, ούτε καν προσπαθούμε. Ο πρόεδρος της Επιτροπής μίλησε για το 2020. Ήδη γνωρίζουμε ότι δεν θα επιτύχουμε τους στόχους, όπως και τους στόχους της Λισαβόνας που δεν επιτυγχάνουμε. Και βέβαια, αποτυγχάνουμε. Ο κύριος Ντόλ ήταν πεπισμένος ε, ότι δεν θέλουμε δεσμευτικούς ε, στόχους. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν είναι έτοιμα να εκπληρώσουν τους στόχους για το 2020, ιδιαίτερα για το περιβάλλον και για την ενέργεια και θα περάσουμε σε αυτό αργότερα. Χρειάζεται δράση και χρειάζεται δράση σύντομα. Η Τραπεζική Ένωση, ο κύριος Σόιμπλε είπε ότι δεν είναι υπέρ της διακυβερνητικής μεθόδου. Προτείνει όμως κάτι το οποίο είναι σαφώ διακυβερνητική μέθοδο, Μα δεν είναι σοβαρά αυτά. Ή είστε υπέρ είτε είστε κατά. Μην προτείνετε κάτι για το οποίο λέτε ότι δεν είστε υπέρ. Δεν είναι έξυπνη πολιτική αυτή. Πραγματική καταπολέμηση τη φοροδιαφυγής, όπω ήδη ανέφερα. Αυτό θα ήταν καλό. Αν την επόμενη εβδομάδα έρθει το Συμβούλιο και μα πει τώρα είμαστε έτοιμοι να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή, θα ήταν πολύ καλό, αλλά δεν το βλέπω. Και πιο δίκαιη κατανομή εισοδήματο βεβαίω, που θα έδινε περισσότερα χρήματα σε αυτού που θα μπορούσαν να τα δαπανίσουν εμφανίσουν και να δημιουργήσουν νέε θέσει απασχόληση, ιδίω πράσινε θέσει απασχόληση. Την περασμένη εβδομάδα η ομάδα μα έκανε μια εξαιρετική συνεδρίαση με τον Ζώσεφ Σίγκλη και άλλου και είδαμε ότι δεν υπάρχει ε, ε, εναλλακτική λύση ε, για τη λιτότητα υπάρχει εναλλακτική λύση της ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Αυτό θέλουμε να επιτύχουμε και αυτό θα πρέπει να επιδιώξει και το Συμβούλιο και η Επιτροπή για να μπορέσουμε να επιτύχουμε και τους στόχους του 2020 για το κλίμα ή τους στόχους του 2030, ό,τι και αν είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Η πολιτική για το περιβάλλον και για το κλίμα μπορεί να επιτευχθεί μόνο με λογική πράσινη ανάπτυξη. Αυτό ζητάμε και ελπίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα μπορέσει το Συμβούλιο για μια φορά να δώσει μια θετική απάντηση στους πολίτες της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σβόμποντα. Εκ μέρους των φιλελευθέρων το λόγο έχει ο κύριος Φερχόφστατ. Ε, ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η τελευταία διάσκεψη κορυφής, το τελευταίο συμβούλιο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές και είναι μια καλή στιγμή για να αξιολογήσουμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Κάνουμε ένα απολογισμό τι έγινε και τι δεν κάναμε και ποιο είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών μας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θέλω να πω ότι τα τελευταία πέντε χρόνια κύριε Μπαρόσο ήταν ε, βέβαια μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, χρέος, κρίση που ξεκίνησε στην Ελλάδα το Δεκέμβριο του 2009. Έχουμε την ε, Αραβική Άνοιξη με πολύ σημαντικά γεγονότα εκεί. Με τους Αμερικανούς φίλους μας έχουμε την υπόθεση κατασκοπίας που συνεχίζεται και για την ε, οποία πρέπει να προβλέψουμε νέα νομοθεσία όσο γίνεται πιο γρήγορα και έχουμε και βαθιά κρίση σήμερα στην Κρυμαία. Θα θυμόσαστε τον ψυχροπόλεμο, βέβαια. Λοιπόν, ήταν μια ταραγμένη εποχή αυτή η τελευταία πενταετία. Πρέπει όμως να είμαστε ε, ειλικρινεί. Γίνανε και πολλά πράγματα από το 2008, από τότε που άρχισε δηλαδή η οικονομική κρίση. Έχουμε τεράστιο νέο δημοσιονομικό κανονισμό μετά από την πρωτοβουλία του Επιτρόπου Μπαρνιέ. Έχουμε οδηγίε σήμερα για την εξηγέση των τραπεζών, για την εκαθάρισή τους. Έχουμε διάφορα προγράμματα στήριξης, δημοσιονομικά μέσα εργαλεία, οδηγίε για την κατάχρηση αγορών. Έχουμε κανονισμό για τους οργανισμούς ε, πιστοληπτικής ικανότητας, κεφαλαίκέ απαιτήσεις κλπ. κλπ. Πολλά έχουν γίνει λοιπόν για την οικονομική διακυβέρνηση και πολλά έχουν γίνει επίσης και χάρη στον συνάδελφο Ρεν όσον αφορά στο σύμφωνο σταθερότητας που επιτέλου εφαρμόζεται. Δεν εφαρμοζόταν πάντα κατά το παρελθόν. Τέλος, έχουμε και θετικά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γιατί χάρη στον κύριο Ντράγκη έπεσε εξάρτηση από τις αγορές. Η πίεση βέβαια δυστυχώς στους πολιτικούς επίσης ε, μειώθηκε. Όμως κατόπιν τούτων είναι αναγκαίο να πούμε την αλήθεια στους πολίτες της Ευρώπης. Δεν έχει τελειώσει η κρίση. Δεν είναι επειδή δεν έχουμε πια ύφεση έληξε και η περίοδος κρίσης και έχουμε μπει σε ανάπτυξη. Όχι, έχουμε μπει σε μία περίοδο που θα λέγαμε οικονομικής ε, σταθερότητας ανάμεσα στο 0 και το 2% με τεράστια ανεργία όμως όπως την ξέρουμε στην Ευρώπη σήμερα. Και αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί λείπουν δύο στοιχεία. Ο Χάινες Βόποντα έκανε τη σύγκριση ανάμεσα στις Ηνωμένε Πολιτείε και την Ευρώπη, τις επιδόσεις μας. Γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Πρώτα απ' όλα γιατί εκείνοι έλυσαν το τραπεζικό τους πρόβλημα. Ενώ εμεί είμαστε ακόμα στη μέση μιας τραπεζικής κρίσης. Δεν έχουμε δημιουργήσει ακόμα το σύστημα εκείνο το οποίο μπορεί να μεταφέρει τα χρήματα από τις τράπεζες στην πραγματική οικονομία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μια μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα, για παράδειγμα, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει επιτόκια 7, 8, 9 και 10 για να κάνει επενδύσεις. Το ίδιο ισχύει και στην Ιταλία δεν θα υπάρξει ανάκαμψη αν πρώτα απ' όλα δεν δημιουργήσουμε μια πραγματική τραπεζική ένωση. Και ο τριμερής διάλογος σήμερα πρέπει να δείξει και να ακολουθήσει τα όσα χθε αποφάσισε το Κοφίν, που δεν ξέρω βέβαια και αν αποφάσισε κάτι τελικά. Τι άλλο χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε και μια ευρωπαϊκή σύγκληση, μια τέτοια πολιτική, μια νέα οικονομική πολιτική. Απέτυχε η ατζέντα της Λισαβόνας του 2020 επίσης, γιατί, γιατί δεν ήταν δεσμευτικά όλα αυτά. Αν έχετε ένα ενιαίο νόμισμα, χρειάζεστε και περισσότερη σύγκληση και περισσότερο δεσμευτική, οικονομική, στρατηγική μεταξύ των διαφόρων μερών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος κάτι εντελώς διαφορετικό. Πιστεύω επίσης ότι την τελευταία αυτή η πενταετία, κύριε Πρόεδρε, είδαμε να μην υπάρχει ενότητα στην πολιτική μας και το βλέπουμε και σήμερα όσον αφορά την Ουκρανία. Δεν υπάρχει ενότητα δηλαδή στην εξωτερική μας πολιτική και δεν υπάρχει θάρρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα είναι δίπλα μας, είναι η γειτονιά μας. Μιλάμε για την Ουκρανία που ουσιαστικά είναι ευρωπαϊκή χώρα. Αν πάτε στην Οδέσα, στο Κίεβο, βλέπετε ότι είσαστε στην Ευρώπη. Και τι κάνουμε? Βλέπουμε την τραγωδία στην Κρυμαία και δεν υπάρχει σοβαρή στρατηγική από τη δικιά μας την πλευρά, ενώ ότι χρειαζόμαστε, που κατά τη γνώμη μου πρέπει να βασίζεται σε διάφορα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα μια κοινή ενεργειακή πολιτική. Ο κύριος Βότσον το είπε. Χρειαζόμαστε δεσμευτικούς στόχους. Είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε μια πραγματική ενεργειακή πολιτική. Έπειτα, χρειάζονται πραγματικέ κυρώσει σε βάρο τη Ρωσία. Σε βάρο του βρώμικου χρήματο που έρχεται από τη Ρωσία και επενδύεται στη Γερμανία, στο Λονδίνο, στη, στα μεσητικά, στι οικοδομέ, στη Γαλλία κλπ. κλπ. Αυτό χρειαζόμαστε. Αλλιώ τελείωσε. Game is over. Θα υπάρξει νέα σύγκρουση για χρόνια. Έπειτα, ευρωπαϊκή η ηγεσία. Δεν πέρασε και πολύ καιρό που οι Ρώσοι ηγέτες από το 90 και μετά δεν είναι έτοιμοι να δεχτούν την ακαιρεότητα των ε, επιμέρους ε, περιφερειών που αποτελούσαν τη Σοβιετική Ένωση πριν. Και το ίδιο συμβαίνει και με την Κρυμαία τώρα. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε είναι να έχουμε θάρρος και να κάνουμε αυτό το οποίο επιβάλλεται και στην Κρυμαία σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φερχόφσετ. Εκ μέρους των Πρασίνων η κυρία Χάρμς έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Μπαρόζο, Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό αν αυτή η τελευταία σύνοδος κορυφής στην οποία προετοιμάζεται, αν θα μπορούσε να αποτελέσει και ένα απολογισμό. Γιατί συχνά τα τελευταία χρόνια ακούμε από την Επιτροπή ότι αντιμετωπίζουμε την κρίση και στο τέλος ε, της δεύτερης ε, θητείας σας ως Πρόεδρου της Επιτροπής έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που χαρακτηρίζεται από πολλές διαιρέσεις βορρά, νότου, ανωτέρων, κατωτέρων στρωμάτων της κοινωνίας και σε μεγάλο βαθμό χειρότερη από ό,τι πριν από πέντε χρόνια και πολύ χειρότερη από ό,τι πριν από δέκα χρόνια. Και θα μπορούσατε να εξηγήσετε τι πήγε στραβά. Θα ήταν ε, χρήσιμο να μας δώσετε ένα τέτοιο απολογισμό. Τώρα θα ήθελα να επικεντρωθώ στην συζήτηση για το κλίμα και την πολιτική ενέργειας και την μελλοντική ικανότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ήδη άκουσα από συναδέλφους πόσο πολύπλοκο είναι το να έχουμε φιλόδοξους στόχους ε, για το κλίμα και για την ενέργεια. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Γερμανία είναι ε, μια χώρα που θα μπορούσαμε να την παρομοιάσουμε με βιομηχανική έρημο. Η οικονομία ε, ε, στη Γερμανία δεν είναι πλέον ανταγωνιστική όσον αφορά τους στόχους για το κλίμα μην, μην γελάτε, δεν μπορούμε να γελάμε γιατί γίνεται μια ανόητη ερμηνεία των διατάξεων για το κλίμα και αυτό οφείλεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική. Επί μια θητεία κύριε Μπαρόζο, ως πρόεδρος της Επιτροπής ε, ε, αναφέρεται δημοσίως ότι είναι φιλόδοξη η στόχη με το Σταύρο Δήμο από την Ελλάδα και με, τον Άντερ Σπίμπαλξ από την Λετωνία. Σε αυτή τη θητεία τους ε, άλλους επιτρόπους, με τον επίτροπο Έτιγκερ, προσπαθήσατε οτιδήποτε είχε δημιουργηθεί να το καταστρέψετε και με αυτούς τους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια που παρουσίασε η δική σας επιτροπή, φτάσατε στο χειρότερο σημείο της διεθνούς πολιτικής για το κλίμα και για ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ο χειρότερος δυνατός. Είναι πραγματικά ε, ε, ε, γελία η κατάσταση και αν δούμε το ε, αν κοιτάξουμε προς Ανατολάς βλέπουμε ότι είναι παράλογη η κατάσταση. Πώς μπορείτε να δικαιολογήσετε αυτή την κατάσταση θα πρέπει σύντομα και μόνο σε αυτό το Συμβούλιο μπορεί να γίνει, θα πρέπει να αναλάβετε την ευθύνη και να διορθώσετε ε, αυτά τα οποία έχετε κάνει για το κλίμα και για την πολιτική. Διαφορετικά στο Παρίσι δεν θα μπορέσουμε να έχουμε καμία επιτυχία, δεν θα γίνει αυτή η διάσκεψη. Με τους στόχους που θέσατε απομακρυνθήκατε από, δύο, ε, από το στόχο του, των δύο βαθμών. Ένα στόχος ε, που είχαμε θεωρήσει ότι από εκεί και πέρα είναι καταστροφικές οι εξελίξεις του κλίματος. Και με τους ε, φιλόδοξους στόχους σας για την προστασία του κλίματος νομίζετε ότι μπορείτε να συνδέσετε την βιομηχανική καινοτομία. Από τις αντιπαραθέσεις στην Κρυμαία και με τη Ρωσία, τι διδασκόμεθα. Τι διδασκόμεθα από την κατάσταση στο νότο, στην Νότια Μεσόγειο. Ότι χρειαζόμαστε ενεργειακή επάρκεια και, ενεργειακούς, ε, και επάρκεια πόρων αλλά ε, εκεί όπου καταπιέζονται άνθρωποι ε, πρέπει η ενέργεια και η επάρκεια, η ενεργειακή επάρκεια και η επάρκεια των πόρων να είναι κεντρικό σημείο της ε, πολιτικής μας. Αυτό από το οποίο εσείς έχετε απομακρυνθεί με την πολιτική σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Χάμς Εκ μέρους του ECR, ο κύριος Ζαραντήλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η χώρα μου προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 10 χρόνια, εδώ και 10 χρόνια. Προσχωρήσαμε με μια μεγάλη ορμή, όμως τώρα βλέπουμε ότι στην τσεχική δημοκρατία δεν υπάρχει εμπιστοσύνη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανέρχεται σε ένα 34%. Είναι ένα πολύ χαμηλό ποσοστό. Και αναρωτιέμαι ποια είναι η αιτία. Ε, ένα παλιό ε, τσεχικό έργο που έφερε τον τίτλο «Πού έκανα λάθος η σύντροφη» με οδήγησε να σκεφτώ ε, ποια είναι και τα δικά μας σφάλματα. Βεβαίως, χάνουμε ΜΜΕ, χάνουμε τα πάντα, γιατί λέμε υποστηρίζουμε τις ΜΜΕ, αλλά τις στραγγαλίζουμε παράλληλα γιατί υπάρχει τρομακτική γραφειοκρατία αλλά στη δική σας δεκαετή θητεία, κύριε Μπαρόζο, δυστυχώς το άχθος της ε, γραφειοκρατίας υπερπολαπλασιάστηκε. Οι πολιτικές υπέρ του κλίματος ήταν ένα μεγάλο φιάσκο. Και το δικό σας διευθυντήριο το λέει αυτό. Είχαμε μία αύξηση κατά 20% των τιμολογίων ηλεκτρισμού. Αύξηση κατά 17% των τιμολογίων ηλεκτρισμού για τις επιχειρήσεις. Και γιατί έγιναν όλα αυτά εξαιτίας της δικής σας πολιτικής ε, για το κλίμα. Ως προς την υποστήριξη των ανανεώσιμων, στο ίδιο οδήγησαν μιλώντας ε, για το 2020 και το 30 και τη μείωση των εκπομπών κατά 40%, τι κάνουμε, τραβάμε το χαλί κάτω από τα πόδια μας. Και τώρα βεβαίως ε, δίνεται μεγάλη μάχη για την ε, Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και τα πολιτικά κόμματα διαλέγουν τους υποψηφίους τους, κάτι το οποίο αντιβαίνει στο γράμμα της συνθήκης. Θα δούμε ποια θα είναι η έκβαση των ευρωπαϊκών εκλογών. Ο κύριος Φερχόφστατ δεν είναι γνωστός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αλλάξουμε τα δεδομένα. Διαφορετικά δεν θα επιτελεστεί ε, καμία πρόοδο. Και τώρα η κυρία Τσίμα, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπαρόζο, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα ασχοληθείτε σίγουρα με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και θα τονίσετε πόσο θετικά είναι τα αποτελέσματα. Είμαστε λίγο πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές και θα ήταν αφελές να περιμένουμε ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα ζητήσουν ε, κάποια σαφήνεια και θα προσπαθήσουν να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Η δική μου πολιτική ομάδα επανειλημμένα ε, έχει ε, τονίσει ότι πρέπει να εξαγαγούμε κάποια διδάγματα από τη διαχείριση της κρίσης τα θύματα της κρίσης ε, δεν έχουν καμία σχέση με την κερδοσκοπία των χρηματαγορών και με την ε, ε, φοροδιαφυγή. Αυτοί όμως υποφέρουν τις συνέπειες. Και τα θύματα της κρίσης δεν νιώθουν την ανάκαμψη της οικονομίας. Αυτό δείχνει πόσο μεγάλες είναι οι κοινωνικές και οι οικονομικές ανισότητες μειώνονται δραστικά οι κρατικοί προϋπολογισμοί εις βάρος αυτών των θυμάτων της κρίσης. Το 2013 η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της, Γερμανίας είχε εξαγωγικό πλεόνασμα 199 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο πλεόνασμα στην ιστορία της Γερμανίας. Ο Επιτρόπος Ρεν το ανέφερε αυτό και είπε ταυτόχρονα ότι γίνονται πολύ λίγες επενδύσεις στη Γερμανία. Ο ρόλος της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι αντίστοιχο με το ρόλο της ε, ποδοσφαιρικής ομάδας ε, της Bayern Βαβαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι κάνει η Bayern στο γερμανικό πρωτάθλημα κάνει και η Γερμανία στην Ευρώπη. Η Bayern ε, είχε ως πρόεδρο ε, κάποιον ο οποίος ε, δικάζεται τώρα για φοροδιαφυγή 27,8 εκατομμυρίων ευρώ από εκεί πέρα, μόνο αλαζονικές δηλώσεις για το πώς μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί μπορούμε να εκφέρουμε. Ε, παρόμοια εκφράζονται και η κυρία Μέρκελ και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σόιμπλε. Η γερμανική συνταγή ισχύει μόνο για τη γερμανική οικονομία και μάλιστα μόνο βράχυπρόθεσμα. Αν δεν αλλάξει κάτι, πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει η δαμόκλειο σπάθη της επόμενης ευρωπαϊκής κρίσης. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου κράτη υψηλές με υψηλό δανεισμό απειλούνται από μακροοικονομική εποπτεία. Γιατί η Γερμανία είχε τεθεί υπό μακροοικονομική εποπτεία. Θα μπορούσαμε να διδαχθούμε από αυτά τα οποία συμβαίνουν. Η διάσκεψη κορυφής θα ασχοληθεί και με την πρόταση της Επιτροπής για τους στόχους για το κλίμα 2020-2030. Με τρόμο ε, διαπίστωσα ότι ε, τα κράτη-μέλη δεν έχουν ε, φιλόδοξους στόχους πλέον και δεν υπάρχει καμία αποτελεσματικότητα η οποία επιζητείται από πλευράς της Επιτροπής. Και είναι τραγικό αυτό, διότι Αυτές είναι παγκόσμιες προκλήσεις και αν δεν μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να τις αντιμετωπίσουμε, αν δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ελάχιστα πλαίσια και κοινωνικά και περιβαλλοντικά προς όφελος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Τσίμε, ο κύριος Φαράτζο εκ ε, του EFD. Ευχαριστώ πολύ η σημερινή ατμόσφαιρα, ακόμη και για το υψηλό επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ιδιαίτερα φορτισμένη. Έχουμε τον κύριο Μπαρόζο και έχουμε μεγάλη συμμετοχή. Τα τελευταία πέντε χρόνια, ε, εγώ είμαι εδώ 15 χρόνια, τα τελευταία πέντε χρόνια κάτι έχει αλλάξει. Καταραίει το ευρωπαϊκό όνειρο. Καταραίει. Στι πρώτε γραμμέ υπάρχουν κάποιοι μανιακοί που θεωρούν ότι ακόμη μπορούμε να τι ονομάζουμε οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Ευρώπη, αλλά οι περισσότεροι ευρωβουλευτέ εδώ, ε, ναι, δουλειά θέλουν, επανεκλογή θέλουν, ο ενθουσιασμός για το ευρωπαϊκό όνειρο πεθαίνει. Και γιατί, διότι έχετε κάνει δύο μεγάλα λάθη. Το πρώτο σφάλμα είναι ότι επεκτείνεται την Ευρωζώνη. Καλά θα ήταν αν ήταν μόνο η Γερμανία και λίγε βορειοευρωπαϊκέ χώρε. Αλλά το να βάλετε και τη Μεσόγειο μέσα στην Ευρωζώνη ήταν καταστροφή. Και το δεύτερο σφάλμα ήταν ότι ε, ε, επιτρέψατε την ελεύθερη διακίνηση ε, προσώπων στην Νότια και Ανατολική Ευρώπη. Είμαστε μια ήπειρο με μετανάστευση. Τώρα έχουμε 4.000 μετανάστες την εβδομάδα που έρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και μένουν ένα χρόνο ή και παραπάνω. Και αυτή είναι η πραγματικότητα που πλήττει τους πολίτες. Δεν λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από οικονομικής πλευράς και το να ανοίξουμε το δρόμο στη μετανάστευση αλλάζει την κοινωνία μας με τρόπο που οι πολίτες δεν το επιθυμούν. Ακούω τα οικονομικά τα οποία αναφέρεται κύριε Μπαρόζο. Είπατε ε, βιομηχανική επανάσταση στην Ευρώπη. Καλό ακούγεται αυτό ε, και σχετική νομοθεσία. Πολύ ενθαρρυντικό και αυτό. Και μετά λέτε ότι πρέπει να επιτύχουμε του στόχου μα για την αλλαγή του κλίματο. Ε, οι Αμερικανοί έχουν επιλέξει το σχιστολιθικό αέριο και μείωσαν τις τιμέ. Οι Κινέζοι βγάζουν κάρβουνο και δεν μπορούμε να του φτάσουμε γιατί ξεκινάνε δύο εργοστάσια παραγωγή ενέργεια κάθε εβδομάδα. Αυτά καταστρέφουν τι θέσει απασχόληση στην Ευρώπη και οι εκλογείς δεν έχουν έχουν θέσεις απασχόλησης και σε λίγες ε, μέρες θα χρειαστεί να δώσουν την ψήφο τους. Ελπίζω ότι στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι πιο συνταρακτικά τα νέα από ό,τι ακούσαμε σήμερα. Ευχαριστούμε. Μία γαλάζια κάρτα από την κυρία Σινκλέρ. Κυρία Σινκλέρ. Σε ποιον απευθύνεται η ερώτηση σας, κυρία Σινκλέρ. Στον κύριο Φαράτζ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Φαράτζ, με την ανεργία που είναι πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, Πιστεύετε κύριε Φαράτζ ότι είναι σωστή χρήση των χρημάτων ε, των ε, φορολογουμένων ε, να δίνετε απασχόληση όχι μόνο στην γυναίκα σας, στην Σαν, αλλά και στην πρώην ερωμένη σας. Έτσι θα πανάτε σωστά τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Θέλετε να απαντήσετε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να απαντήσω, λέει ο κύριος Φαράτζ. Κύριε Μαγκίνες. Um, Ελπίζω τη δικιά μου την ερώτηση να την απαντήσετε κύριε Φαρέντς. Μιλάτε για ενθουσιασμό στην πολιτική. Με κάθε σεβασμό. Εγώ δεν θέλω ενθουσιασμό. Θέλω κόσμο που δουλεύει. Μπορείτε να δεσμευτείτε ότι θα παραμείνετε εδώ και θα ακούσετε τις απαντήσεις που θα σας δώσουν αυτοί που θα παραμείνουν εδώ, γιατί η πρακτική σας κατά το παρελθόν είναι να σηκώνεστε και να φεύγετε. Μιλάτε για τον ενθουσιασμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέτε ότι μειώνεται. Ο ενθουσιασμός για το UKIP μειώνεται. Um, Αν ήταν μια κανονική ερώτηση θα απαντούσα, αλλά ο ευρωσκεπτικισμός αυξάνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς εδώ ούτε και πιο μανιακοί που πιστεύουν στο οικοδόμημα δεν τον θυζητούν αυτό. Φαίνεται από τη δεξιά, την αριστερά, το κέντρο, παντού. Και ο λόγος, είσαστε από την Ιρλανδία, το ξέρετε καλύτερα από οποιοδήποτε, ο λόγος είναι ότι κανείς ποτέ δεν έδωσε συνένεση για μια ευρωπαϊκή πολιτική συνένεση. Οι Γάλλοι, οι Ολλανδοί απέρριψαν το σύνταγμα το οποίο μεταμορφώθηκε στην ε, συνθήκη. Οι Ιρλανδοί το απέρριψαν. Οπότε δεν μπορείτε να πείτε ότι υπάρχει λαϊκή στήριξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση της Ευρώπης. Μπορεί να το πιστεύουν η κυρία Μέρκλου, ο κύριος Μπαρόσο, αλλά οι λαοί της Ευρώπης όχι. Ο κύριος Μπρόνς. Ευχαριστώ. Για να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε, μερικές φορές πρέπει να έχουμε διαφορετικές πηγές και να τις βάλουμε μαζί. Λοιπόν, η ατζέντα αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που σημαίνει ότι η Κομισιόν εποπτεύει και ελέγχει τα μεταρρυθμιστικά προγράμματα στην αγορά. Και μιλάμε για βιομηχανικό ανταγωνισμό, ότι θέλουμε ε, ανταγωνιστικότητα που θα δημιουργήσει απασχόληση. Ας πάμε όμως πίσω σε μια συνάντηση ΕΚΟΦΗΝ 16 Φεβρουαρίου του 2012 για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο τότε θα διαπιστώσουμε ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, είπανε, στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα μηχανισμούς για τη ρύθμιση των μισθών ώστε να προσαρμοστεί το εργασιακό κόστος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μια οικονομία με υψηλούς μισθούς και με την λογική της ε, παγκοσμιοποίησης πρέπει να μειώσει τους μισθούς για να μπορεί να ανταγωνιστεί τις αναδυόμενες οικονομίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιαννάκου, εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι είναι το τελευταίο Συμβούλιο πρώτων Ευρωπαϊκών Εκλογών και γι' αυτό έχει ιδιαίτερη και τεράστια σημασία. Και βέβαια το περιεχόμενό του, η ατζέντα του, δίνει έμφαση στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, το οποίο απαιτέλεσε μια πολύ θετική διαδικασία που αποφασίστηκε τα τελευταία χρόνια στην ουσία κλείνουμε πέντε χρόνια μιας οικονομικής κρίσης πάρα πολύ σκληρής για την οποία ελήφθησαν συγκεκριμένα μέτρα και έγιναν συγκεκριμένες ενέργειες. το σύμφωνο ανάπτυξης και σταθερότητας θεωρείται υποχρεωτικό πλέον και δεν παραβιάζεται ούτε από μεγάλες ούτε από μικρές χώρες και τεράστιες αλλαγές συνέβησαν στην περιοχή μας στον περίγυρο της ευρώπης μπόρεσε αυτές τις αλλαγές είτε την αραβική άνοιξη είτε όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στις παλιές σοβιετικές δημοκρατίες να τα αντιμετωπίσει από κοινού η ευρωπαϊκή ένωση. όχι. παρά τις προσπάθειες ο διακυβερνητισμός εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό στοιχείο λειτουργίας και τη βασική μέθοδο εργασίας στην ουσία. ο τρίλογος για συγκεκριμένα θέματα καθυστερεί αφόρητα και συγκρούσεις μεταξύ των κρατών μελών γίνονται για ελάχιστα συμφέροντα κάτι που φυσικά δεν συνέβαινε στην αρχή της δημιουργίας της ευρωπαϊκής ένωσης. ωστόσο η ένωση αυτή προσφέροντας 50 χρόνια ευημερίας και ειρήνης σε όλους τους πολίτες τους έδωσε το δικαίωμα και την πολυτέλεια να είναι πολύ κριτικοί απέναντί της. πρέπει να τονίσουμε τα αρνητικά αλλά και συγχρόνως τα θετικά και να σημειώσουμε κύριε πρόεδρε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανταπόκριση στα ζητήματα που ετέθησαν από τους συναδέλφους πραγματική αν δεν υπάρξει μια πραγματική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια πραγματική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Επομένως μας χρειάζεται μια διαφορετική Ευρώπη. Αυτό που λένε ορισμένοι περισσότερη Ευρώπη, αλλά διαφορετική, όπου θα ξεκαθαριστεί τι απομένει στα κράτη-μέλη και τι ανάκειται σε ευρωπαϊκή πραγματική διακυβέρνηση η οποία μπορεί να κάνει τις αλλαγές που χρειάζονται είτε στη φορολογία είτε να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή είτε να συντονίσει τα δικαιοπρακτικά συστήματα είτε να λειτουργήσει ως πραγματικά ενιαίος χώρος. αυτό πρέπει να είναι το ζήτημα που θα απασχολήσει το επόμενο συμβούλιο μετά τις εκλογές στις οποίες εγώ προσωπικά ελπίζω ο ευρωσκεπτικισμός όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως από τον κύριο farage να μην έχει ιδιαίτερα σημαντική θέση. Ευχαριστούμε κύριε Γιαννάκου. Κυρία Φεραίρα, εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών. Η Τραπεζική Ένωση ίσως είναι το βασικότερο κληροδότημα της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για την επανοικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την κρίση. Μπορεί να επέλθει συμφωνία με το Συμβούλιο πριν από το τέλος της θητείας, εάν υπάρχει πολιτική βούληση. Η συνεισφορά της Επιτροπής ήταν ύψιστη για το κείμενο νομοθετικού περιεχομένου. Θα θέλαμε όμως η Επιτροπή να ήταν πιο αποφασιστική στην ε, υποστήριξη αυτού του προγράμματος προγράμματος. Ε, κατά τον τριμερή διάλογο του ΕΚΟΦΗΝ, ο κύριος Στουρνάρας μαζί με τον κύριο Ντάισελ Μπλουμ ε, βρέθηκαν δίπλα-δίπλα, κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερα συμβολικό που σημαίνει ότι θα υποβληθούν σοβαρές προτάσεις για να φτάσουμε σε συνένεση θεωρώ ότι δεν μπορούμε να μειώνουμε την ποιότητα των κειμένων μας επειδή είναι κατεπήγοντος χαρακτήρα. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η εντολή διαπραγμάτευσης ε, είναι συγκεκριμένη. Έχουμε μία τραπεζική ένωση που δεν θα δέχεται τα τραπεζικά παιχνίδια. Θα πρέπει οι φορολογούμενοι να μην πληγούν. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το προφίλ επισφάλειας των τραπεζών και να δούμε αν καταδικάζονται ή όχι. Και αυτό για να είμαστε αξιόπιστοι. Το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει στις ε, διαπραγματεύσεις, διότι μία κακή συμφωνία θα πλήξει την ίδια την Τραπεζική Ένωση. Είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε το νομοθετικό κείμενο. Θα πρέπει όμως να είμαστε ιδιαίτερα ε, υπεύθυνοι και αναμένουμε τις εξελίξεις. Θεωρούμε ότι τα νόμιμα ευρωπαϊκά συμφέροντα θα υπερισχύσουν όλων ναι. των άλλων. Κυρία Πρασίνων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι η πρώτη συζήτηση για το κλίμα και την ενέργεια ενώπιση του 2020 και είναι τώρα που πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι για τις κλιματικές αλλαγές, γιατί πρέπει να περιοριστούν εκπομπές, κάτι που χρειάζεται ακόμα περισσότερο σήμερα από ότι ποτέ για να μην ε, ανέβει η θερμοκρασία τόσο πολύ στον πλανήτη. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερο ποσοστό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να ακούσουμε τους επιστήμονες, ε, τα στοιχεία. Οι έρευνες δείχνουν ότι χρειάζονται υψηλή στόχη γιατί έτσι θα μειωθεί και η εξάρτησή μας από τις εισαγωγές και θα μειωθούν οι δαπάνε για την ενέργεια. Δεν είναι δηλαδή μόνο περιβαλλοντικό το επιχείρημα, είναι και οικονομικό. Θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση, πολύ βασικό, κυρίω για του νέου. Χρειαζόμαστε λοιπόν βιώσιμη απασχόληση στον ενεργειακό τομέα. Γνωρίζω από τη δικιά μου περιφέρεια, την Ουαλία, ότι στρέφονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για λύσεις. Πρέπει να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας στον κόσμο ότι θα καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Ζητάω λοιπόν από το Συμβούλιο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Εύανς. Κύριε Σαλβίνη, εκ μέρους των EFT. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχει πεθάνει το ευρώ. Το λένε τα αριθμητικά στοιχεία. Μπορεί να σκοτώσει και την Ευρώπη που γεννήθηκε ε, μετά από μια πολύ καλή ιδέα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την κρίση ε, της αυτοκτονίας των επιχειρηματιών και ούτω καθεξής. Λυπάμαι που ο πρόεδρος Μπαρόζο δεν είχε χρόνο να ακούσει και ορισμένες επικρίσεις. Οι Βρυξέλλες ε, υπερασπίζονται τις πολιεθνικές και τις μεγάλες τράπεζες. Δεν υπερασπιζόμαστε τις μικρές μας τις δικές μας επιχειρήσεις. Η Ινδία, η Αμερική, ο Καναδάς, η Βραζιλία υπερασπίζονται το made in, δηλαδή το δικό του σήμα, ενώ εμείς κατακρεουργούμε χιλιάδες επιχειρήσεις. Άρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να σώσουμε την Ευρώπη, γιατί το ευρώ έχει ήδη πεθάνει. Άρα θα πρέπει να οικοδομήσετε τα πάντα εκ νέου. Ο κύριος Ρόιλ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν υπάρχει πρόοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν είναι τόσο που είναι ανυπέρβλητα. Δεύτερον, υπάρχει πρόβλημα ανάπτυξης και απασχόλησης και γι' αυτό πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Σαφώς υπάρχει βελτίωση και θα πρέπει να φροντίσουμε ε, να αντιμετωπίσουμε την αποβιαμηχανοποίηση στις ευρωπαϊκές χώρες. Μόνο σε πέντε χώρε ανήστε η βιομηχανοποίηση από το 2007. Μόνο εννέα ευρωπαϊκές ε, Βιομηχανίε, ανήσουν στι ισχυρότερε του κόσμου. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με τη βιομηχανία και την ανάπτυξη και αυτό όχι μέσω χορηγήσεων κονδυλίων αλλά μέσω ρυθμιστικού πλαισίου. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο. Δεν έχει νόημα το να θέτουμε όλο και περισσότερου στόχου και να επιβαρύνουμε τη βιομηχανία μα χωρί νόημα. Χρειαζόμαστε έξυπνου στόχου, έξυπνα προγράμματα, κίνητρα για να μπορέσουμε να έχουμε έχουμε έρευνα και καινοτομία, να υποστηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες και το αποτέλεσμα της πολιτικής μέχρι τώρα μπορεί να βελτιωθεί. Χρειάζεται να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας μέχρι τώρα. Πρέπει να προωθήσουμε τη βιομηχανία, χρειαζόμαστε περισσότερα προγράμματα ανταγωνιστικότητας, χρειαζόμαστε ε, ένα υψηλότερο ποσοστό για την βιομηχανία, αυτό που ανέφερε η Επιτροπή για το 20% και η βιομηχανική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βελτιωθεί. Ευχαριστώ πολύ και τώρα εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών ο κ. Γκερέιρο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πριν από λίγα λεπτά μόλις ο κύριος Βόμποντα αναφέρθηκε στο κίνδυνο το νέο συμβούλιο, το νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να έχει τα δύο χαρακτηριστικά που ζημιώνουν περισσότερο και οδηγούν στην ανάδρεια πρώτα απ' όλα να συνεχίσει ως business as usual και δεύτερον να καταλήξει σε έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή, ελάχιστης φιλοδοξίας δηλαδή. Μιλάμε για την ενέργεια. Πριν από λίγες εβδομάδες μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τους στόχους του για το κλίμα. Ενέκρινε επίσης μία προσπάθεια της τάξης του 30% για τις ανανεώσιμες, μείωση 40% των εκπομπών και επάρκεια ενεργειακή της τάξης του 40%. Τι έκανε η Ευρωπαϊκή λοιπόν, Επιτροπή μετά την απόφαση του Κοινοβουλίου υπέβαλε μια πρόταση πολύ λιγότερο φιλόδοξη και όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και χωρίς κανέναν στόχο για την ε, ενεργειακή επάρκεια. Μας λένε ότι το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο πρέπει να περιμένουμε μια νέα πρόταση. Θα είναι τις παραμονές που θα σταματήσει να υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ο κύριος Βαρόσο γνωρίζει, καταλαβαίνει τα ισπανικά, θα καταλάβει και αυτό που λέμε στα ισπανικά ότι ποτέ δεν είναι αργά όταν δεν έχουμε κάνει τίποτα. Τι θα γίνει λοιπόν? Το ατύχημα στη Φουκουσίμα οι νέες τεχνολογίες που είναι όλο πιο αποτελεσματικές, η ανασφάλεια ενεργειακή που έχουμε μετά τα γεγονότα στην Ουκρανία απαιτούν μεγαλύτερη προσπάθεια από τη δικιά μας την πλευρά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για την ενεργειακή απόδοση και για την διασύνδεση. Η ομάδα μου τσακώθηκε για να πετύχει δεσμευτικούς στόχους και πιο φιλόδοξους. Η Γερμανία έχει μια φιλόδοξη ενεργειακή πολιτική και άλλες χώρες όπως η Ισπανία όχι, δυστυχώ. Αντίθετα, καταστρέφουν την προσπάθεια για τι ανώσιμε πηγές ενέργεια και οδηγούνται σε ένα χάο ηλεκτρική ενέργεια που σίγουρα θα αποτρέψει τις επονδύσεις και θα μειώσει τις προσπάθειες ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε κύριε Ο κύριος Λαβία, εκ του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Προεδρεύοντα, Κύριε Επίτροπε, βρισκόμαστε σε μια στιγμή όπου τα μάτια των πολιτών είναι στραμμένα προς τα θεσμικά όργανα. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στις ευρωπαϊκές εκλογές και αυτό που έχει σημασία είναι τι κάναμε μέχρι τώρα και τι θα κάνουμε στο μέλλον. Ό,τι έγινε δεν επαρκεί διότι τα αποτελέσματα είναι ενώπιαν όλων μας. Βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικοί και αποκλίνοντες δείκτες μεταξύ κρατών μελών. Το Εαρινό Συμβούλιο το οποίο ασχολείται με θέματα ανταγωνιστικότητας, σήμερα θα αποφάσισε να ασχοληθεί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το κλίμα και την ενέργεια. Μα αυτά είναι τα μοναδικά θέματα. Δεν πρέπει να εξεύρουμε νέα μέσα και μηχανισμούς. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία για να ενισχύσουμε την ανάπτυξη και χρειαζόμαστε νέα χρηματοοικονομικά μέσα για τις επιχειρήσεις. Οι πόροι είναι πολύ περιορισμένοι. Το Youth Guarantee δεν αρκεί. Ο δείκτης ανεργίας είναι πολύ υψηλός. Και ως προς την Τραπεζική Ένωση βεβαίως είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Θα πρέπει όμως να λειτουργήσουμε μαζί διότι τα επιτόκια είναι πολύ ψηλά. Θα πρέπει να πέσουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σήμερα είναι υπερβολικά ψηλά. Η Μπαχές, μέρος των Σοσιαλδημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση αυτή. Μιλάμε για το τελευταίο Ευρωπαϊκό Ιαρινό Συμβούλιο, οπότε χαίρομαι που έχουμε τη συζήτηση αυτή. Ο πρόεδρος Παρόσο δεν κατάλαβε τελικά σε τι χρησιμεύει ένα αερανό συμβούλιο. Δεν είναι δυνατόν για να εφαρμόζεται ένα ευρωπαϊκό εξάμεινο, ένα εξάμεινο λιτότητας. Δεν μπορεί να χρησιμεύει για ένα ευρωπαϊκό εξάμεινο το οποίο δεν βλέπει τον κοινωνικό κατακαιρματισμό στην Ευρώπη μετά από 10 χρόνια εντολής του κύριου Παρόσο. Δεν μπορεί να είναι ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που λέει ότι χρειάζονται κοινωνικοί δείκτες αλλά τελικά δεν ε, λαμβάνει υπόψη καμία συνέπεια. Δεν μπορεί να είναι ένα ευρωπαϊκό εξάμεινο που πιστεύει ότι οι δείχτες ανάπτυξη είναι ικανοποιητικοί, που θεωρεί ότι η στρατηγική 2020 είναι επιτυχία, ενώ όλοι οι δείχτες είναι στο κόκκινο και κανένας στόχος της στρατηγικής 2020 δεν θα επιτευχθεί. Ήρθε καιρό να αλλάξουμε πλειοψηφία, ήρθε καιρό να αλλάξουμε κομισιόν, ήρθε καιρό να έχουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή στρατηγική που να μα επιτρέψει να έχουμε μια συνολική αντίληψη και να δώσουμε προτεραιότητα στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που να μας επιτρέψει να κάνουμε την απασχόληση μια πραγματική προτεραιότητα. Για όλα αυτά, ο κύριος Μπαρόσο εδώ και 7 χρόνια καθόρισε την ιδέα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ενέργειας. Αλλά βλέπουμε ότι δεν μπόρεσε να την εφαρμόσει τελικά. Σήμερα είμαστε στην καρδιά του ρήγματος αυτού, του ενεργειακού ρήγματος εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που λείπει η ηγεσία μας μιλάει για βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Ναι, αλλά τι έκανε για να βοηθήσει η ενέργεια αυτή να υπάρχει για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Έπρεπε να υπάρχει πολιτική βούληση και ηγετικές ικανότητες για να το πετύχουμε αυτό, για να έχουμε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας που θα γεννήσει απασχόληση παντού στην Ευρώπη. Συνεπώς, χαίρομαι που ίσως μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στα φορολογικά ε, της ενέργειας, στη απουσία του κυρίου Γιούνκερ στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπερές. Εκ μέρους ε, του ΕΛΚ, ο κύριος Οντή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαίρω τον πρόεδρο Μπαρόζο και τον πρόεδρο Βαν Ρόμποη για όσα κάνουν για να ξεκινήσει μια πολιτική σκέψη. Κύριε Μπερέση, απευθυνθείτε στον πρόεδρο τη Γαλλική Δημοκρατία που είναι μέλο ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και που μπορεί και να επηρεάσει τι αποφάσει που λαμβάνονται και όχι στον πρόεδρο Μπαρόζο, ο οποίο εκτελεί αυτά που εμεί αποφασίζουμε. Επίση, λυπάμαι που δεν προβλέπεται και μια διάσκεψη κορυφή τη ευρωζώνη ε, που προβλέπεται από το από το Σύμφωνο Ανταγωνιστικό ε, Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός ε, ε, ο στόχος που έχει τεθεί. Πρέπει όλες οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, λαμβάνουν υπόψη τη βιομηχανική πολιτική. Το ίδιο και την πολιτική ανταγωνιστικότητα. Στην περιοχή του Λιμουζά ακόμη ε, είμαστε υπό το σοκ του ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αρνήθηκε να συγχωνευτούν δύο μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες για να γίνουν μια τεράστια παγκόσμια εταιρεία στον τομέα της ηλεκτρονικής. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και για την εμπορική πολιτική. Ας μην είμαστε είμαστε ε, αφελείς και μιλάμε για την ε, αμοιβαιότητα. Ε, το ίδιο και για την νομισματική πολιτική. Κλείνοντας θέλω να μιλήσω και για τις εκλογές. Οι πολίτες πρέπει να έχουν τον τελευταίο λόγο θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη συζήτηση με πολλά έγγραφα, με τη γνώμη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, με τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενδιάμεση, στρατηγική, ε, ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής 2020 και με τις προοπτικές για τις προσεχείς πολιτικές συζητήσεις για τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές 2016. Κύριε Οντί, έχετε μια ερώτηση από την κυρία Μπεχές. Κυρία Μπεχές. Κύριε Οντί, επιλεκτικά διαβάζετε την επικαιρότητα. Δεν θα σας διαφεύγει ότι ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας πρότεινε σημαντικές πρωτοβουλίες για την ενέργεια και γαλλογερμανική συνεργασία, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες. Αυτό νομίζω ότι συνάδει προς τα όσα εμείς εδώ προτείνουμε. Ο κύριος Οντί. Την ερώτησή σας δεν την, δεν την βλέπω ως ερώτηση. Ναι, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, πράγμα το οποίο δεν το έκανε η κυβέρνησή του πριν από ένα χρόνο, όντως ασχολείται με τη γαλλογερμανική συνεργασία και τον συγχαίρω γι' αυτό. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκιούρκ, εκ μέρους του ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, Η βιομηχανία στην Ευρώπη παίζει σημαντικό ρόλο για την απασχόληση και για την ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Υπήρου στην παγκόσμια οικονομία έχει οπισθοχωρήσει. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και θα πρέπει να φροντίσουμε να ξαναμπούμε στο τρένο της ανάπτυξης. Η κατάσταση της βιομηχανίας χάλιβα είναι ενδεικτική. Η οικονομική κρίση παράλληλα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα, που μερικές φορές ξεχνά την πραγματικότητα, δημιουργεί ένα τεράστιο ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τη βιομηχανία χάλιβα και η ανταγωνιστικότητα παίζει σημαντικό ρόλο ούτως ώστε ε, να έχουμε και την τεχνολογία που απαιτείται και να είμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο σημαντικοί. Πρέπει να φροντίσουμε να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας, διότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία πληρώνει διπλάσια και τριπλάσια τιμή για την ενέργεια σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερα μέτρα σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ράγκελ και πάλι από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το πρώτο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι για μας είναι αποφασιστική σημασία ο τριμερής διάλογος και η μεγάλη όθηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Αφορά την Τραπεζική Ένωση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μία προοπτική ανοίγματο και ευελιξίας για να ανταποκριθούμε στις, να ανταποκριθεί το Συμβούλιο στις θέσεις της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Η, η Πορτογαλική κυβέρνηση υπό τον Πάσο Σκουέλιου ε, ζήτησε να ληφθεί υπόψη η σημασία μιας πραγματικής τραπεζικής ένωσης και όχι ένας διακυβερνητικός κατακαιρματισμός της. Αυτό ακριβώς ανέφεραν ανέφερε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Μάιερ, στα πλαίσια της διάσκεψης του ΕΛΚ. Υπάρχουν χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία που αντιμετωπίζουν μεγάλες ανάγκες και γι' αυτό δεν πρέπει να υφίστανται κυρώσεις από την κατάσταση της χώρας τους. Δεν πρέπει να υφίστανται κυρώσεις οι επιχειρήσεις τους. Θα πρέπει μία επιχείρηση να την χάνει της ίδιας αντιμετώπισης είτε βρίσκεται στην Αθήνα, είτε στη Στοκχόλμη, είτε στη Λισαβόνα, είτε στο Βερολίνο. Ο κύριος Φανινίστελ Ρόι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε το Made in Europe, ό,τι παράγεται στην Ευρώπη, θα έπρεπε να έχει την προτεραιότητα. Υπάρχει γνώση στην Ευρώπη που οδηγεί όμως την παραγωγή σε άλλα μέρη του κόσμου. Εμείς χάνουμε την παραγωγή από τα χέρια μας. Θα έπρεπε να είναι αλλιώ τα πράγματα. Η νέα γενιά, για παράδειγμα, ε, φωτοβολταϊκών, η νέα τεχνολογία πρέπει και να παράγεται και εδώ και μετά να εξάγεται από εδώ. Θα πρέπει δηλαδή να αλλάξει η νοοτροπία μας. Να αλλάξουν οι δομές ε, ορίζοντας 2020 και τα λοιπά, θα πρέπει να υπάρχει διασύνδεση με τη βιομηχανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει κάποια καλά βήματα, ο κύριος Σταγιάννη, ο Επίτροπος Χάν, αλλά πρέπει να προχωρήσουν περισσότερο έχουμε εμπιστοσύνη. Πρέπει να υπάρξουν περισσότερες εγγύσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για πράσινη απασχόληση. Όσον αφορά εμένα, αυτή πρέπει να είναι δεσμευτική στόχη για το μέλλον. Ευχαριστούμε κύριε Βενσερόη. Περνάμε στο Catch the Eye. Ε, ναι, ομιλητέ έχουν ζήσει το λόγο. Αν θέλετε όλοι να κρατήσετε το χρόνο που σας έχει δοθεί, θα μπορέσουμε να ακούσουμε και τους εννέα ομιλητέ. Κύριε Μακίνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να καθίσουμε και να σκεφτούμε ότι όταν συζητάμε τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Προεδρεύων του Συμβουλίου πολύ σωστά αναφέρθηκε στην κατάσταση στην Ουκρανία, θέλω να κάνω μερικά σχόλια για το πού βρισκόμαστε. Κανένας στο σώμα αυτό, σίγουρα όχι από την πλευρά μας, δεν θα έλεγε ότι όλα είναι ρόδινα. Ξέρουμε ότι στην Ιρλανδία πάρα πολλοί άνθρωποι δεν νιώθουν την βελτίωση που θα θέλαμε να δουν. Αλλά πρέπει συγχρόνως να παραδεχτούμε ότι υπάρχει σταθερότητα, ότι υπάρχει ανάπτυξη. Πολύ μικρή βέβαια, πάρα πολύ μικρή, που πρέπει να ενισχυθεί. Στηρίζω πάντως στα σχόλια του κ. Φανίστερόι που λέει ότι πρέπει η παραγωγή να επανέλθει στην Ευρώπη, να μπορούμε να δημιουργήσουμε βιώσιμη απασχόληση εδώ. Τέλος, στην Ιρλανδία οι στόχοι δεν ήταν βιώσιμοι, υπέφερε ο κόσμος, αλλά πρέπει να του δώσουμε ελπίδα. Ευχαριστούμε κυρία Κάλεμπαχ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Κουρκούλα, Αναφέρετε ότι η διάσκεψη κορυφή θα ασχοληθεί με την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, με την ενέργεια και το κλίμα. Διότι όλοι αυτοί οι τομείς θα πρέπει να συνδυάζονται. Κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει απλώς να συνδυάζονται Αντίθετα με τον κύριο Ντόλ, εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμους ε, φιλόδοξους ε, στόχους για να διασφαλίσουμε το μέλλον της Ευρώπης, αλλά ε, χρειαζόμαστε και μια Ευρώπη της ευημερίας για να διασφαλίσουμε θέσεις απασχόλησης και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης. Για να είναι η ενέργεια βιώσιμη θα πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο δεν θα θέτει σε κίνδυνο το μέλλον, τις μελλοντικέ γενιές. Αν δεν είμαστε επαρκείς στις ανάγκες της τωρινής γενιάς όσον αφορά την εκπαίδευση και την απασχόληση, θέτουμε σε κίνδυνο και την τωρινή και τις μελλοντικέ γενιές. Ευχαριστώ η κυρία Μπιλμπάου Παραντιγά. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύοντα, ε, επαναλαμβάνω αυτά που είπε ο δικός μας ε, Λεντακάρη στους υπεύθυνους Ευρωπαίους. Θα πρέπει να υπάρχει συσχετισμός με την άμεση οικονομία. Θα πρέπει να, να διασωθεί η απασχόληση και όχι να διασώζονται μόνο οι τράπεζες. Θα πρέπει να δίνονται πιστώσεις στις επιχειρήσεις, διότι η λύση βρίσκεται στην πραγματική οικονομία, στο ανθρώπινο δυναμικό, στους άνδρες και τις γυναίκες που είναι η μοχλή της πραγματικής οικονομίας. Ναι, στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά με κοινωνική ανάπτυξη. Οι, Κι, οι εργάζονται χωρίς ε, κοινωνική προστασία. Δεν πρέπει να φτάσουμε στα στο ίδιο σημείο. Διαφορετικά δεν είναι βιώσιμος ο κόσμος. Λυπάμαι που αποχώρησε ο κύριος Μπαρόζο, διότι θα ήθελα να διαβιβάσει αυτά που προείπα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο, στη διάσκεψη της Νέας Υόρκης το Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλάμε για θέσει επασχόληση οι Ευρωπαίοι για τις βιομηχανίες θεωρήσαν ότι θα δημιουργήσουμε μέχρι το 2030 50.000 θέσεις απασχόλησης. Μπορούμε να πούμε όχι σε θέσεις απασχόλησης όταν έχουμε 20 εκατομμύρια ανέργους. Ο Επίτροπος Μπαρόζο ανέφερε και τώρα στρέφομαι στον κύριο Ρεν. Χρειαζόμαστε δεσμευτικούς στόχους ε, για το 2020 και 2030 για να έχουμε αυτές τις θέσεις απασχόλησης. Ευχαριστώ κυρία Κρόνμπεργκ, Ο κύριος Πρόεδρε, θα συζητήσουμε σε λίγο για τα περί Ουκρανίας και Ρωσίας. Θέλω να σας πω ότι είχαμε τις πρόλες στην ε, Γεωργία. Σήμερα έχουμε την Ουκρανία, μεθαύριο θα έχουμε τη Μολδαβία. Τι θα γίνει λοιπόν με την ε, πολιτική αυτή τι θα κάνει την επόμενη φορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τι πρέπει να κάνει μάλλον. Να έχει υπόψη ότι η Ουκρανία είναι μια από δια, πιο διαφθορμένε χώρε του κόσμου και γι' αυτό, σε αυτό έχουν να κάνουν και ο κύριο Γιανουκόβιτ και η κυρία Τιμουσέμκο. Άρα λοιπόν και θα δικηθεί σύντομα στο διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Έπειτα, το μόνο που ενδιαφέρει τον Πούτιν είναι η τραπεζική του λογαριασμοί. Συνεπώς οι ολιγάρχες και ο Πούτιν είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε. Και τρίτον, ενεργειακή πολιτική. Πρέπει να αναθεωρηθεί πλήρω η ενεργειακή μα πολιτική και να είμαστε ανεξάρτητοι από το ρωσικό φυσικό αέριο. Τζίπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ θα ήθελα να τονίσω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γνωρίζει την κατάσταση, η κατάσταση στην Ουκρανία και η ενέργεια και το κλίμα από την άλλη πλευρά. Όλα αυτά συμβαδίζουν διότι η ενεργειακή προμήθεια, η ασφάλεια ενεργειακής προμήθειας είναι ύψη της σημασίας και τη βλέπουμε υπό ένα συγκεκριμένο πρίσμα των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας η πολιτική για το κλίμα θα πρέπει να λάβει υπόψη τους ε, μεγάλους ε, παίκτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κινηθεί από μόνη της. Η πολιτική ενέργειας θα πρέπει να οριστεί από τα κράτη-μέλη. Έτσι θα αναζωογονήσουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία και θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Χάσαμε εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 20 εκατομμύρια είναι άνεργοι. Αυτό θα έπρεπε να βρίσκεται επιτάπητος και όχι κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Ταβάτση. Ε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μας ε, ενδιαφέρουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Μας ενδιαφέρουν και τα ενεργειακά δίκτυα που να συμπεριλαμβάνουν όμως πολλά κράτη-μέλη. Για την Ουγγαρία δεν θα υπήρχε άλλη λύση πέραν της διασύνδεσης αυτών των δικτύων, ιδίως αν εκλείψει ο εφοδιασμός από την Ρωσία. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα συνετοί με την ένταση που επικρατεί στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή. αυτή η ένταση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας λόγω Ουκρανίας θα μπορούσε να επηρεάσει την εύθευστη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βάγκελ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, πιστεύω ότι τα γεγονότα στην Ουκρανία αλλά και άλλες παγωμένες συγκρούσεις στην Κρυμαία και αλλού σημαίνουν ότι ανοίγει μια νέα περιοχή κρίσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, συνεπώς, θα πρέπει να καθίσει να σκεφτεί τι γίνεται με την κοινή εξωτερική μας πολιτική. Μπορεί να αντικατασταθεί από ad hoc ταξίδια υπουργών που πάνε στο Κίεβο και που τελικά καταλήγουν σε σκανδαλώδη αποτελέσματα όπως η τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στη Λέιδη Άστον και τον Εστονό Πρωθυπουργό ή από παρεμβάσεις υπουργών ε, τη στιγμή που δεν κρατάνε ούτε καν 24 ώρες. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να δείξει τι είναι ικανή να κάνει, λύνοντας τέτοιες παγωμένες συγκρούσεις αντί να δημιουργεί νέες. Χρειαζόμαστε μια κοινή εξωτερική πολιτική και οι ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων πρέπει να φροντίσουν και να δώσουν ένα σαφές μήνυμα για το πώς πρέπει να είναι η πολιτική αυτή. Ευχαριστούμε. Ο τελευταίος αυτό τον γύρο ΚΑΤΣΤΙΑΙ είναι η κυρία Άννα Γκόμες. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, πώς μπορούμε να έχουμε μία αξιόπιστη βιομηχανική πολιτική, εμπορική πολιτική ανταγωνισμού, εάν το Συμβούλιο και η Επιτροπή παραβλέπουν την φορολόγηση στα κράτη-μέλη και το σκάνδαλο της φοροδιαφυγής. Πρόσφατα η γερουσία των ΗΠΑ διενέργησε ακροάσεις και έδειξε ότι οι ελβετικές τράπεζες συμμετέχουν στην φοροδιαφυγή Αμερικανών πολιτών. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Ευρωπαίους ενώ ζητούμε φορολόγηση από τους φτωχούς και τη ε, μεσαία τάξη, οι ζάπλουτοι χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα το οποίο είναι απαράδεκτο. Άρα τι κάνουν οι Επίτροποι και το Συμβούλιο για να θέσουν τέρμα σε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστούμε Άννα έληξε η διαδικασία Catch the Eye και θα δώσουμε το λόγο στον Αντιπρόεδρο Όλη Ρεν για να αντιδράσει στις διάφορες παρεμβάσεις. Κύριε Ρεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για την τόσο σοβαρή και ουσιαστική συζήτηση που είχαμε για τα θέματα που έχουν να κάνουν με το επερχόμενο Ιαρινό Συμβούλιο. Πρέπει να σας πω ότι είχα την τάση να σημειώσω κάποια σημεία και να σηκώσω κι εγώ την μπλε μου κάρτα για να ρωτήσω όχι μόνο τον κύριο Φαράς αλλά και άλλους για τα επιχειρήματά τους. Αλλά τέλος πάντων δεν τη βρήκα εδώ την μπλε κάρτα οπότε δεν τα έκανα. Οπότε θα αναφερθώ σε διάφορα σημεία στα συμπεράσματά μου. Θα θυμόσαστε ότι στην προηγούμενη Ολομέλεια συζητήσαμε για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο επί μακρό. Και είχαμε και τις ε, προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη και βλέπουμε ότι η ανάκαμψη κερδίζει έδαφος. Και οδήγησε περισσότερη εγχώρια ζήτηση και γίνεται πιο ευρωστή στις περισσότερες χώρες μέλη, ακόμα και στις πιο ευάλωτες. Την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύτηκε ανάλυση και συμπεράσματα μετά από τις οικονομικές επισκοπήσεις που έγιναν για τις 27 οικονομίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δείχνουν ότι υπάρχει πρόοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζει τις οικονομικές δυσκολίες, αλλά ότι η πρόοδος αυτή είναι άνηση και μερικές ε, φορές πρέπει να ενισχυθεί πολύ περισσότερο, ιδιαίτερα σε τομείς όπως είναι η απασχόληση, όπου η ανεργία σε πολλές χώρες αποτελεί μάστιγα. Τα κράτη-μέλη, λοιπόν, πρέπει να στηρίξουν επικοδομητική συνεργασία προκειμένου να σταθεροποιηθεί η ανάκαμψη και να υπάρξουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Το στοιχείο κλειδί πάντως όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις χώρες της Ευρωζώνης είναι και συνεχίζει το ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη στην Ιταλία και στη Γαλλία να ενισχύσουν τις οικονομικές τους μεταρρυθμίσεις υπέρ της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης ενώ συγχρόνω πρέπει να ενισχυθεί η εσωτερική ζήτηση, η εγχώρια ζήτηση και να υπάρξουν επενδύσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στην Γερμανία. Όλα αυτά είναι συμπληρωματικά βέβαια και με μια τέτοια στρατηγική μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όσο γίνεται καλύτερα την αηφόρο ανάπτυξη και την δημιουργία απασχόληση στην Ευρώπη. Και αυτό ακριβώς είναι που χρειαζόμαστε αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Συνεπώς, είναι ζωτική σημασία να συνεχίσουμε με τις μεταρρυθμίσεις σε όλες τις χώρες μέλη. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με οικονομικές μεταρρυθμίσεις, έχει να κάνει με ένα μεγάλο εύρος μεταρρυθμίσεων βασικών για να ανακτηθεί ανταγωνιστικότητα και να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Έχει να κάνει επίσης με τη φοροδιαφυγή. Αναφέρθηκε εδώ πολλοί από εσά αναφερθήκατε στην φοροδιαφυγή, η κυρία Γκόμεση ήταν η τελευταία. Πράγματι είναι σημαντικό όχι μόνο για να είμαστε οικονομικά πιο αποτελεσματικοί, να συλλέγονται φόροι, αλλά για να υπάρχει και κοινωνική δικαιοσύνη και ο κόσμος να βλέπει ότι δεν πληρώνουν μόνο ε, μερικοί, αλλά ότι το βάρος ε, καταμερίζεται ισότιμα μεταξύ όλων. Αναφερθήκατε επίσης στον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Πρέπει να πω ότι προσβλέπω σε συνεργασία με τον τεο συναδελφό μου και φίλο μου, Jean-Claude Juncker, προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στο Λουξεμβούργο, κάτι το οποίο είναι πολύ βασικό για τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαίρεται για τα θέματα που έχει το Ερεινό Συμβούλιο, που είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και η ενέργεια και οι κλιματικές αλλαγές. Όντως πρέπει να καταπολεμηθούν οι κλιματικές αλλαγές. Άκουσα πολύ προσεκτικά την κυρία Χάρμς για παράδειγμα και πρέπει να σας πω με κάθε σεβασμό ότι οι πράσινοι δεν εξυπηρετούν την Ευρώπη υποτιμώντας την σημαντική συνεισφορά μας και τον ηγετικό μας ρόλο παγκοσμίω όσον αφορά τι κλιματικέ αλλαγέ. Γιατί είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται από πάρα πολλέ αρχές. Από τον Αλγκόρ, από τον Νικολα Στέρν και τον Μπάνκι Μουν. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό εμείς οι ίδιοι να μην αυτό πυρπολούμεθα. Ο ο Ακιμούν, και άλλοι το έχουν πει ότι κάνουμε πολλά στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Το αναγνωρίζουν αυτό, αναγνωρίζουν τον ηγετικό ρόλο δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν. Η πράσινη ανάπτυξη πρέπει να γίνει το βασικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητάς μας γιατί θα βοηθήσει και στην οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση. Η Ευρώπη πρέπει να κάνει πολλά πράγματα. μεταξύ άλλων και στην κλιματική και ενεργειακή πολιτική και στην ενιαία αγορά και στη νέα βιομηχανική μας πολιτική. Η Ευρώπη πρέπει να καθορίσει τους στόχους και να δώσει όθηση. Όμως οι χώρες μέλη θα αποφασίσουν για την εφαρμογή και θα επιλέξουν τα ίδια ποια είναι τα δυνατά του σημεία και μετά θα λειτουργήσει η αγορά και οι επιχειρήσεις θα βρουν τις πιο καινοτόμες λύσεις στον τομέα, για παράδειγμα, της βιοοικονομίας και της καθαρής ενέργειας. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας, από ό,τι φαίνεται, είναι να έχουμε έναν στόχο για την μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και ένα πρόγραμμα καταπολέμησης των εκπομπών. Αυτό σε συνδυασμό με οικονομικές μεταρρυθμίσεις θα ανακτηθεί η ανταγωνιστικότητα, θα προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη και θα βγούμε από την κρίση με μια πιο δυνατή οικονομία και πιο βιώσιμη από ό,τι κατά το παρελθόν. Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με το εξής ακολουθήσει συζήτηση για την Ουκρανία μετά από αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα. Θέλω να υπογραμμίσω λοιπόν ότι η Ευρώπη στηρίζει το δικαίωμα των Ουκρανών να αποφασίσουν για το μέλλον τους, για τον ευρωπαϊκό τους προσανατολισμό. Θέλουμε να βοηθήσουμε την Ουκρανία να σταθεροποιήσει την κατάσταση, να έχει ασφάλεια, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξουν και οι προϋποθέσεις για οικονομική σταθεροποίηση και οικονομική ανάπτυξη. Γι' αυτό το σκοπό την προηγούμενη εβδομάδα Είχαμε μια ερευνητική αποστολή στην Ουκρανία προκειμένου να βοηθήσουμε τις προπτικές για οικονομική βοήθεια προς τη χώρα. Τώρα αναλύουμε τα αποτελέσματα της αποστολής αυτής και είμαστε σε στενή επαφή με το Κίεβο και την αποστολή του Εθνούς Νομισματικού Ταμείου εκεί. Την προηγούμενη εβδομάδα επίσης Είχαμε και το πολιτέ πακέτο αρρωγή για την Ουκρανία που ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προηγουμένη. Μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ μπορούν σύντομα και σταδιακά να δοθούν υπό τη μορφή δανείων και μακροοικονομικής αρρωγής. Αυτά επιπλέον από τα 600 εκατομμύρια ευρώ ένα δισεκατομμύριο δηλαδή συνολικά θα εκταμιευθεί μόλις υπάρξει πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Επιτόπου. Και βέβαια θα εξαρτηθεί, είναι υπό την προπόθεση, μεταρρυθμίσεων που πρέπει να κάνει η Ουκρανία ώστε να γίνει πιο ανθεκτική, πιο εύρωστη και να μπορεί να βοηθήσει έτσι καλύτερα τους Ουκρανούς εφόσον βέβαια είναι σοβαρή για την καταπολέμηση της διαφθοράς εκεί. Στην Ουκρανία είναι αλήθεια ότι πρέπει σιγά σιγά να υιοθετηθεί το πακέτο αυτό και ελπίζω να έχετε στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έγκριση του οικονομικού αυτού πακέτου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε πίτροπε Ρεν. Τώρα το λόγο έχει εκ μέρους του Συμβουλίου ο Υπουργός Κούρκουλας. Ευχαριστώ πολύ αγαπητά μέλη. Σας ευχαριστώ για αυτή την άκρο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ακούσαμε ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων για όλα τα θέματα τα οποία είναι αλληλένδετα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτά τα ζητήματα συμβαδίζουν. Μας ενδιαφέρουν και οι εξελίξεις στην Ουκρανία και θα πρέπει να αντιδράσουμε σοβαρά και με συντονισμό. Αυτό δεν είναι κάτι το ξεχωριστό από τα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Πολύ τονίσατε την κοινωνική πτυχή. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι ένα θέμα ζωτικής σημασίας και βασίζεται ε, στην κοινωνική οικονομία της αγοράς. Εάν υπάρχει ανισορροπία μεταξύ στοιχεία της αγοράς και στοιχείων της αγοράς και κοινωνικών στοιχείων, ε, βασίζεται στο γεγονός ότι δεν ε, έχουν προωθήσει τα ζητήματα, τα ζητήματα αυτά τα κράτη-μέλη. Η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη υπάρχει, αλλά είναι ευάλωτη. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε με την διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και με μεγάλη σοβαρότητα. Είναι ένα πολύ σοβαρό μέσον για να συνεχίσουμε με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη. Όπως τονίστηκε από πολλά μέλη, έχει επιτελεστεί πρόοδος στο θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης Επίσης αναφερθήκατε σε οικονομικο-χρηματικούς μηχανισμούς στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάκαμψης στην Τραπεζική Ένωση που είναι ζωτικής σημασίας και στην Ελληνική Προεδρία φιλοδοξούμε να εγκριθεί ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης. θα διενεργηθεί ένας τριμερής διάλογος στις 3 σήμερα στο Ταρασβούργο με τους Υπουργούς Οικονομικών και τον Πρόεδρο του Eurogroup. Έχουμε αναλάβει μία νέα εντολή και ας ελπίσουμε να είναι μία ε, σταθερή βάση για να επιτευχθεί ένα συντονισμός. Διαφορετικά θα πρέπει να αναπέμψουμε το ζήτημα στις κυβερνήσεις ζητώντας ε, μία ευέλικτη εντολή. Αυτό είναι θέμα αξιοπιστίας της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κούρκουλα για την ε, παρέμβαση του Συμβουλίου. Κλείνει η συζήτηση αυτού του πολύ σημαντικού ζητήματος της ημερήσιας διάταξης. Το επόμενο θέμα είναι οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το θέμα που φέρει τον τίτλο «Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία».